Bien. Mes Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είμαστε εδώ σε αυτή την επιβλητική αίθουσα για την συνεδρίασή μας τη σημερινή. Πριν κηρύξω την έναρξη των εργασιών μας, επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τις ευχές μου για μια εξαίρετη νέα χρονιά 2018 τόσο προσωπικά με τους φίλους σας, στην οικογένειά σας όσο βέβαια και επαγγελματικά για όλα τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις εργασίες της δικιάς μας ειδική Επιτροπής για την Τρομοκρατία εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ήρθατε. Πρώτα απ' όλα, ημερήσια διάταξη, έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να σας ζητήσω να την εγκρίνουμε. Υπάρχει αντίρρηση. Όχι. Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν η ημερήσια διάταξη. Και περνώ τώρα στις ανακοινώσεις της Προεδρού. Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερο από την προηγούμενη συνεδρίασή μας που έλαβε χώρα τις παραμονές των χριστουγεννιάτικων διακοπών. Οπότε έτσι θα περάσω δίχως άλλο στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με τον Μάικλ Οφλάχερτη που είναι ο Διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν σήμερα το απόγευμα υποδεχόμαστε εδώ τον Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που ήρθε ε, όλος ιδιαίτερος για μας από την Αυστρία ε, και από την Αυστραλία από ό,τι κατάλαβα και που ήρθε να μας ε, μιλήσει και να συζητήσει κυρίως με την Επιτροπή μας για τα θέματα που μας απασχολούν. Θα θυμόσαστε αγαπητοί συνάδελφοι ότι συμφωνήσαμε από την αρχή της εντολής της Επιτροπής μας, κατά τη σύνταξή της δηλαδή, αλλά και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια των προηγούμενων συνεδριάσεων της Επιτροπής μας, συμφωνήσαμε λοιπόν για την διάσταση αυτή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και για το πόσο σημαντική είναι αυτή και ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία για την διάσταση αυτή και να τη λαμβάνουμε υπόψη μας σε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή μας, κάθε φορά δηλαδή που συζητάμε κάτι εδώ. Εξάλλου, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Θεμελιδών Δικαιωμάτων, όπω γνωρίζετε, πάντα υπογράμμιζε τη σημασία που έχει αυτή η προσέγγιση ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάθε φορά που συζητάμε για θέματα ασφάλεια και ότι η διάσταση αυτή των θεμελιωδιών δικαιωμάτων μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία, τα θύματα της τρομοκρατίας, να τα βοηθήσουμε και από την άλλη να μπορέσουμε πιο σωστά να λάβουμε υπόψη μας ό,τι έχει να κάνει με ανταλλαγή πληροφοριών εδώ. Κάθε φορά λοιπόν σε όλα αυτά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και το έργο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που έχει δουλέψει πάρα πολύ και όσον αφορά τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, αλλά και όσον αφορά την ασφάλεια στα εσωτερικά και εξωτερικά μα σύνορα. Επίσης και όσον αφορά το σεβασμό του ιδιωτικού βίου και την προστασία των ε, πληροφοριών που έχουν να κάνουν με τον ιδιωτικό βίο, τα προσωπικά δεδομένα. Υπάρχει ένα εξαιρετικό έγγραφο το οποίο δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2017, σωστά, από τον οργανισμό σας για τα θέματα αυτά η γραμματεία ίσως θα μπορούσε στα πρακτικά τη σημερινή μας συνεδρίαση να βάλει και το αυτό. Οπότε, κύριε ο αν συμφωνείτε, παρουσιάστε μας παρακαλώ τα κύρια θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το σεβασμό των θεμελιδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, που είναι και θέμα της δικιάς μας Επιτροπής. Οπότε θα σας δώσω το λόγο για 15-20 λεπτά το πολύ και στη συνέχεια, όπως είπαμε, θα περάσουμε στις ερωτήσεις και τις απαντήσεις. Οπότε οι συνάδελφοι, και συγγνώμη αν χρειαστεί να σας κόβω, θα πρέπει να τηρήσουν το χρόνο τους. Δηλαδή ένα λεπτό ο καθένας για την ερώτησή του, έτσι ώστε να μπορέσει και ο Διευθυντής να μας απαντήσει. Σε πέντε λεφτά περίπου, εκεί μπορεί να είμαι πιο ελαστική. Στόχος είναι να μπορέσουμε να έχουμε διάλογο, συζήτηση μεταξύ μας και να απαντηθούν όλες οι ερωτήσεις των συναδέρφων. Σας ευχαριστούμε που δεχτήκατε λοιπόν αυτή τη διαδικασία και χωρίς άλλη καθυστέρηση σας δίνω και το λόγο κύριο Φλάιρτη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω που καλέσατε τον Ευρωπαϊκό Οργασμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων να έρθει σήμερα και να συζητήσει μαζί σας. Σας συγχαίρω επίσης και για το έργο σας στην Ειδική Επιτροπή για την Τρομοκρατία. Διότι μια ασφαλής Ευρώπη είναι πολύ βασική και για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Οι τρομοκρατικές ενέργειες αποτελούν απειλή για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Και ιδιαίτερα για το δικαίωμα στη ζωή, που είναι και το πιο βασικό δικαίωμα. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να πω ότι έχουν ε, ιδιαίτερη σημασία σήμερα, είναι πιο επίκαιρα από ποτέ, ακριβώς επειδή κλείνουν τρία χρόνια από την επίθεση που έγινε στο Παρίσι. Προσπαθούμε λοιπόν να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία με διάφορους τρόπους, λαμβάνοντα όμω πάντα υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα. Πρέπει κανεί ακούμε συχνά σήμερα, να διαλέξει περισσότερη ασφάλεια ή περισσότερο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όμως δεν είναι αυτή η περισσοτερο σεβασμο των ανθρωπινων δικαιωματων ομω Δεν είναι αλήθεια ότι έχει εχει κανει να διαλέξει. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ασφάλεια αποτελούν ένα δίδυμο, ένα τάντεμ και πάνε χέρι-χέρι. Το ένα δεν αποτελεί εμπόδιο για το άλλο. Αντίθετα, μόνο προστατεύοντα τα θεμελιώδη δικαιώματα μπορούμε να έχουμε περισσότερη ασφάλεια. Έτσι λοιπόν υπάρχουν τα Ενωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουν τα σταγματικές υποχρεώσεις που ισχύουν πάντα, ακόμα και όταν έχουμε να κάνουμε με τις προκλήσεις που μας δημιουργεί η τρομοκρατία. Χρειάζεται ελαστικότητα προκειμένου να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προκλήσεις αυτής. Ο περιορισμός των δικαιωμάτων δεν βοηθάει. Πρέπει πάντα να τηρεί την νομιμότητα, η αναγκαιότητα, η αναλογικότητα και να τηρούμε και την αρχή της μη διάκρισης. Από τις έρευνες που έχει κάνει ο οργανισμός μας, και από την εμπειρία που έχω εγώ, στην οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, φαίνεται ότι οι θεμελιώδη δικαιώματα δεν πρέπει να τα βλέπουμε σαν ένα εμπόδιο προκειμένου για να πετύχουμε μια ασφαλή κοινωνία μέσα στην οποία να μπορούν να μεγαλώσουν τα παιδιά μας με ασφάλεια. Σεβόμενοι τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρώντα τις αρχές που πριν ανέφερα, δημιουργούμε και μια βιώσιμη ατμόσφαιρα, ένα βιώσιμο κλίμα μέσα στις χώρες μέλη. Σήμερα λοιπόν δεν μπορώ βέβαια να καλύψω όλα τα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που έχουν να κάνουν με το έργο σας. Οπότε αυτό που θα κάνω είναι ότι θα αναφερθώ στις έρευνες που έχει κάνει ο οργανισμός μας και θα επικεντρωθώ σε τρεις τομείς. Πρώτα απ' όλα, πώς θα αποφύγουμε τη ριζοσπαστικοποίηση. Δεύτερον, στα θέματα της ασφάλειας και της μετανάστευσης. Και το τρίτο έχει να κάνει με το πώ εφαρμόζεται η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατά τη τρομοκρατία σε εθνικό επίπεδο. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έρχομαι στη ριζοσπαστικοποίηση. Καλωσορίζουμε τι προσπάθειε της Επιτροπής σας προκειμένου να αποφεύγεται η ριζοσπαστικοποίηση και προκειμένου να αποφεύγονται όλες οι πηγές τρομοκρατίας. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Θεμελιδών Δικαιωμάτων συγκεντρώνει στοιχεία προκειμένου να σας βοηθήσει. Τον Εύρη, για παράδειγμα, που μας πέρασε, δημοσιεύσαμε τη μεγαλύτερη ανάλυση που έγινε ποτέ βάσει των εμπειριών που έχουμε από τους Ευρωπαίους μουσουλμάνους για να διαπιστώσουμε ποιες, ε, ποια είναι τα προφίλ, ποια είναι, ποιες είναι οι πατέντες που ακολουθούν. Με 10.500 ανθρώπους σε 15 χώρες μέλη έγινε η ανάλυση αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν μετανάστες, είτε πρώτης είτε δεύτερης γενιάς, αλλά η μισή από αυτούς είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Οπότε θα αρχίσω με κάτι που ίσω δεν περιμένετε. Με τα καλά νέα από την ανάλυση αυτή, από την έρευνα αυτή όσον αφορά τη στρατηγική μα κατά τη ριζοσπαστικοποίησης. Και αυτό είναι ότι υπάρχουν υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών των κοινοτήτων ε, Ευρωπαίων Μουσουλμάνων, ότι δηλαδή εμπιστεύονται του Ευρωπαϊκού θεσμού περισσότερο από ότι ο γενικό πληθυσμό. 81% λοιπόν εξέφρασαν την προσέγγιση τους ε, στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και 60% είπαν ότι είναι ιδιαίτερα, ε, αισθάνονται ιδιαίτερα κοντά σε αυτούς. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο για τις κοινωνίες μας. Πρέπει όμως συγχρόνως να είμαστε προσεκτικοί, γιατί τα επίπεδα του σεβασμού αυτού, στα πλαίσια των εμπειριών που έχουμε με διακρίσεις και οχλήσεις, πρέπει ε, να μας κάνουν να βρούμε τρόπους να συνεχίσουμε με την εμπιστοσύνη αυτή και όχι να καταστραφεί αυτή. Συνεπώς, ο οργανισμός μας πιστεύει, κατέληξε δηλαδή στο συμπέρασμα από την ανάλυση αυτή αλλά και από άλλες έρευνες, ότι η καταπολέμηση της ριζοσπαστικοποίησης απαιτεί μεταξύ άλλων και την καταπολέμηση του μοντέλου που ακολουθούν, δηλαδή να αντιμετωπιστούν τα παράδεκτα επίπεδα διακρίσεων που υπάρχουν στους χώρους εργασίας, στην εκπαίδευση, και σε πολλά και διάφορα πλαίσια όπου χρειάζεται ακόμα πιο έντονη καταπολέμηση της ρητορική μίσους. Στα πλαίσια αυτά και πάλι βάσει των εργασιών του Ευρωπαϊκού Οργασμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να σας πω ότι ακούμε πολλά για το ποια είναι η στρατηγική που λειτουργεί καλύτερα για την ένταξη των ανθρώπων αυτών και ποια είναι η στρατηγική που έχει αποτύχει. Πράγματα τα οποία νομίζω ότι ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή σας για να δούμε πώς θα καταπολεμηθεί η ριζοσπαστικοποίηση. Συνεπώς, από τις έρευνες που κάναμε και που δημοσιεύτηκαν πριν από ένα χρόνο, έχω να σας πω εξής. Πρώτον, πρέπει να βρεθούμε πιο κοντά με στρατηγικές τοπικές ένταξεις που λειτουργούν καλύτερα από ότι εκείνες που γίνονται σε κεντρικό επίπεδο. Να δουλεύουμε δηλαδή στους Δήμους συγκεκριμένα. Δεύτερον, κάτι προφανές αλλά που πρέπει να το πούμε γιατί δεν γίνεται αρκετά, οι στρατηγικές ένταξεις απαιτούν ανάπτυξη σε διαβούλευση με τις ομάδες των ανθρώπων που θέλουμε να ενταχθούν, αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό. Πρέπει δηλαδή να γνωριστούν μεταξύ τους όλες αυτές οι πλευρές. Και τρίτον, πρέπει να εντάξουμε και προσεγγίσεις που έχουν να κάνουν με το φύλλο. Γιατί πολλές φορές οι προσέγγιση μας είναι ουδέτερη όσον αφορά το φύλλο. Κάτι το οποίο δεν είναι πάντα θετικό. Η ουδετερότητα αυτή σημαίνει ότι αποκλείουμε τις εμπειρίες των γυναικών που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας αν θέλουμε να πετύχουμε. Και τέλος οι εργασίες μας δείχνουν ότι ο ρόλος των στρατηγικών ένταξης δεν υπόκειται επαρκώς σε τακτική αξιολόγηση. Πολλές ε, χώρες μέλη κάνουν βέβαια πιο καλά τη δουλειά, δηλαδή μαθαίνουν από τις ε, εμπειρίες ε, τις δικές τους και των άλλων. Τώρα όλα αυτά, την ανάλυση αυτή και τα αποτελέσματα των ερευνών μας αποτελούν μέρος της συνεισφορά μας στην ομάδα υψηλού επίπεδου της Επιτροπής για την ριζοσπαστικοποίηση, όπου συμμετέχουμε. Προσπαθήσαμε με τον τρόπο αυτό να εντοπίσουμε και να πούμε ναι, η ριζοσπαστικοποίηση φυσικά και χρειάζεται την προσέγγιση της ασφάλειας, αλλά συγχρόνως αυτό σημαίνει και μια δέσμευση από την πλευρά μας να συνεργαστούμε με τις διάφορες κοινότητες, να αντιμετωπίσουμε ε, τα προβλήματα τα κοινωνικά και τα οικονομικά που αντιμετωπίζουν συχνά οι κοινότητες αυτές και να λάβουμε υπόψη μας τα προβλήματα των ανθρώπων που ζουν επί τόπου. Και να σας πω για τη δικιά μου εμπειρία που ήμουνα υπεύθυνο σε μια Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πριν, ότι η προσέγγιση αυτή της ασφάλειας, αν συνδυαστεί με την κοινοτική προσέγγιση, καταλήγει σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. Έτσι αποφεύγεται η ζωστικοποίηση. Και ήμουνα στην Βόρεια Ιρλανδία ε, επίτροπο σε μια τέτοια επιτροπή και πρέπει να σας πω ότι είδα εντυπωσιακά αποτελέσματα ακριβώς μετά την σύγκρουση που είχαμε στη Βόρεια Ιρλανδία και πώς καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα τραύματα του παρελθόντος. Οι επόμενοι τρει τομεί έχουν να κάνουν με τα θέματα τη ασφάλεια και τη μετανάστευση από του τρει τομεί ο επόμενο. Ξεκινώ λοιπόν με τα όσα είπε ο Επίτροπο Τζούλιαν Κίνγκ στην Επιτροπή σα πρόσφατα, όταν σα κάλεσε να αποφύγετε να αποφύγετε τη σύγχυση των θεμάτων της μετανάστευσης με τα μελήματα τα σχετικά με την ασφάλεια. Και είναι πολύ θεμητό αυτό, δηλαδή σας επεσήμανε πως το να έρθουν σε αντιπαράθεση τα θέματα αυτά εξυπηρετεί το παιχνίδι των εξτρεμιστών. Και πολύ σωστά το λέει, συμπληρώνω ταυτόχρονα ότι πέραν του ότι εξυπηρετεί το παιχνίδι των εξτρεμιστών, υποβιβάζει την αναγκαία προστασία των ανθρωπινών δικαιωμάτων των αθώων αυτών, στου οποίου συγκαταλέγονται βέβαια και τα παιδιά θα συμπληρώσω. Χωρί βέβαια επουδενή, κυρία Πρόεδρε, να θέλω να υποδείξω ότι θα πρέπει να ε, απαλληφθεί, να λησμονηθεί το θέμα της ασφάλειας στο μεταναστευτικό. Όχι, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούμε να ε, αναγνωρίζουμε τη μετανάστευση ως πηγή της τρομοκρατίας. Αλλά πρέπει να ακολουθήσουμε την προσέγγιση του Julian King. Και αυτό σημαίνει ταυτόχρονα και σημαντική δουλειά για την ε, οργάνωση, την υπηρεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κάνει πολύ σημαντική μελέτη και στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της μετανάστευσης, ιδιαίτερα θεμελιώδη δικαιώματα στο χώρο αυτό με την μελέτη που κάναμε πρόσφατα ταυτόχρονα και σε συνεργασία με την ε, υψηλού επίπεδου Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συλλογή δεδομένων στα ε, σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ιδιαίτερα για το θέμα αυτό της διαλειτουργικότητας, που γνωρίζω βεβαίως ότι ε, είναι από τα κύρια ζητήματα που σας ενδιαφέρουν, θέλω να πω τα εξής και ξεκινώ επισημένοντας ότι η υπηρεσία θεμελιωδών δικαιωμάτων χρειάζεται την διαλειτουργικότητα, προσφέρει τη διαλειτουργικότητα που είναι απαραίτητη για διάφορους λόγους, για την ασφάλεια αλλά και για την ενίσχυση των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Επί παραδείγματι, η αναζήτηση παιδιών των οποίων έχουν χαθεί τα ίχνη. Με τη διαλειτουργικότητα θα βελτιωθεί ασφαλώς η ε, αναζήτηση και η εξέβρεση των παιδιών αυτών. Η διαλειτουργικότητα βεβαίως πρέπει και μπορεί να εξασφαλιστεί κατά τρόπον ώστε να εξυπηρετείται και ο σκοπός της προστασίας των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Έτσι λοιπόν στη δική μας συνεισφορά σε αυτήν την ομάδα υψηλού επίπεδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπογραμμίζουμε τα εξής πολύ σημαντικά. Πρώτον, η αρχή του περιορισμού του στόχου, του σκοπού. Στη διαλειτουργικότητα, παραδείγματι, σας καλούμε με ιδιαίτερη προσοχή να εξετάζετε την διαφύλαξη των ορίων εξυπηρέτηση ενό στόχου. Δηλαδή τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται θα πρέπει να εξυπηρετούν μόνο το στόχο για τον οποίο συλλέγονται. Ταυτόχρονα, ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε το γεγονό ότι η συλλογή δεδομένων με τα συστήματα αυτά θα πρέπει να γίνεται με τρόπο επακριβή, γιατί είναι πολλά τα σφάλματα και το εντοπίζουμε πολλέ φορέ στη δουλειά μα. Επί παραδείγματι, κάναμε πρόσφατα συνεντεύξεις με ε, υπαλλήλους που εργάζονται στα σύνορα, οι οποίοι εντοπίζουν, όπως μας είπαν συχνά, σφάλματα στην εισαγωγή δεδομένων, στις βάσεις δεδομένων κατά τη διάρκεια της δουλειάς τους, στο σύστημα θεώρησης διαβατηρίων, είναι παραδείγματι, αλλά και στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν. Σφάλματα τα οποία βεβαίως ε, οδηγούν σε πολλά προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά γεννούν και πολλά ζητήματα ασφάλειας γιατί ένα μη ακριβές σύστημα δεδομένων, ένα ανεπαρκές ή ατελές σύστημα δεν μπορεί να υποστηρίξει και το πλαίσιο της ασφάλειας. Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη έχετε λάβει προτάσεις σε σχέση με τη διαλειτουργικότητα, κατόπιν βέβαια του έργου της ομάδας υψηλού επίπεδου των εμπειρογνωμόνων, που σε μεγάλο βαθμό λαμβάνουν υπόψη και τις δικές μας προτάσεις και χαιρόμαστε γι' αυτό. Βεβαίω οι προτάσει αυτέ συμπεριλαμβάνουν και στοιχεία τα οποία δεν έχουν τύχει επαρκού προσοχή σε επίπεδο ομάδα εμπειρογνωμόνων, που όμω έχουν σημαντικέ συνέπειε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα ιδιαίτερα να επισημάνω τα εξή δύο κεφάλαια που φαντάζομαι θα πρέπει να σα απασχολήσουν. Πρώτον, προτάσει σχετικέ με την ικανότητα τη διαλειτουργικότητα να αναγνωρίσει πολλαπλέ ταυτότητε ενό μεμονωμένου ατόμου πρώτον και δεύτερον, η διαλειτουργικότητα μπορεί να εντοπίσει υπηκόους τρίτων κρατών για, και παραθέτω από το έγγραφο της Επιτροπής, λόγους ε, δημόσιας πολιτικής ή δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας ε, ασφάλειας σε σχέση με το διεθνές δίκαιο. Χωρίς να θέλω να επεκταθώ περισσότερο, θέλω να επισημάνω στην Επιτροπή σας ότι δεν έχουν τύχει επαρκούς προσοχής τα σημεία αυτά σε επίπεδο Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων υψηλού επίπεδου. Και γι' αυτό θέλει ιδιαίτερη έχει ιδιαίτερη σημασία η δική σας ε, δουλειά και προσοχή. Και τρίτον, ε, Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ στις ε, στην εφαρμογή από τι εθνικέ αρχέ αρχές της νομοθεσίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και εδώ θα επισημάνω το εξή. Έχει πραγματοποιήσει το Κοινοβούλιο σα ιδιαίτερα σημαντική δουλειά ω προ την ε, ε, εφαρμογή τη οδηγία για την καταπολέμηση τρομοκρατία που υιοθετήθηκε πέρσι. Πέραν όμω αυτή τη καλή δουλειά, τα πραγματικά αποτελέσματα τη εφαρμογή αυτή τη οδηγίας θα εξαρτηθούν από την εθνική υλοποίηση ε, ιδιαίτερα στου τομεί εκείνου που επιτρέπουν περιθώριο ερμηνεία σε εθνικό επίπεδο, όπω ε, τα σημεία που έχουν να κάνουν με το χαρακτηρισμό αδικημάτων ως προς την υπόθελψη ή την υποκίνηση τρομοκρατικών ενεργειών. Οι διασφαλιστικές δικλείδες για τα θεμελιώδη δικαιώματα που αναφέρονται στην οδηγία αυτή λοιπόν πρέπει να είναι ε, σημείο και κομμάτι αναπόσπαστο της εθνικής νομοθεσίας για την υλοποίηση της οδηγίας. Επίσης, η υποστήριξη η βοήθεια που θα προσφερθεί στα θύματα της τρομοκρατίας έχει πολύ μεγάλη σημασία. Πολύ συχνά λησμονούνται, δεν την χάνουν επαρκούς προσοχής τα θύματα αυτά ως ομάδα πληθυσμού και αυτό το έχω παρατηρήσει και από τη δουλειά μου στη Βορεια Ιρλανδία. Παραμελείται λοιπόν η, το σύνολο των αναγκών τους, ε, δεν δίνεται επαρκής προσοχή στα θύματα της τρομοκρατίας. Τα στοιχεία της οδηγίας που αναφέρονται στα δικαιώματα των θυμάτων πρέπει να μεταφερθούν σε εθνικό δίκαιο κατά τρόπο ορθό. Και σε αυτό θέλω ιδιαίτερα να επιμείνω. Έτσι κυρίες και κύριοι, για να ολοκληρώσω, θα ήθελα εκ μέρους της υπηρεσίας μας να εκφράσω και πάλι ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη για τη δουλειά σας, για την προσέγγισή σας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτή σας η δουλειά για μας και πιστεύουμε ότι κατά την εκτέλεση αυτού του έργου έχει πολύ μεγάλη σημασία να, εντοπιστεί, να αναγνωριστεί ότι δεν υπάρχει σχέση ανταγωνισμού μεταξύ ανθρωπινών δικαιωμάτων και ε, καταπολέμηση τρομοκρατία. Αντιθέτω, συστήματα τα οποία σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βελτιώσουν σημαντικά και τα συστήματα τα σχετικά με την ασφάλεια. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να ε, δηλώσω την διαρκή μας υποστήριξη και βέβαια με την παρουσία μου εδώ και το υλικό το οποίο σας φέρνουμε και στην αίθουσα αυτήν, αλλά ταυτόχρονα και με την διαθεσιμότητα για απαντήσεις σε οποιαδήποτε παρατήρησή σας ή για, σε ανάγκες για περαιτέρω αναλύσεις. Είμαστε πάντα στη θέση σας. Ευχαριστώ πολύ. Euh, σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση, κύριε Φιντά. Ήταν πυκνή, εξαιρετικά επίκαιρη και σίγουρα ε, τροφοδοτεί τη συζήτηση και τα ερωτηματικά των συναδέλφων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κατερίνα Κινίτσι και η Μπίρκη Τσίπελ μετά, ο Ζόφρε, Βανότεν. Ας αρχίσουμε. Ένα λεπτό έκαστος για κάθε ερώτηση παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Οφλαερτή για την ε, τοποθέτηση σας για άλλη μια φορά με πληρέστατο αλλά και συνοπτικό τρόπο μας παρουσιάσατε όλα τα ζητήματα και την πρόταση την οποία με χαρά υποδέχομαι του συνδυασμού της ε, καταπολέμησης τρομοκρατίας με το σεβασμό των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω τις επισημάνσεις σας και για την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, στην οποία και εγώ εργάστηκα. Βεβαίως θα πρέπει στη συνέχεια όλα αυτά να μεταφραστούν σε συγκεκριμένες ε, δράσεις, ε, πέραν των υποδείξεων δηλαδή της οδηγίας, να δούμε συγκεκριμένα τι γίνεται στο εθνικό δίκαιο κατά τη μεταφορά. Και εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ζήτημα της αντιμετώπισης της ρίζοσπαστικοποίησης. Για τη ρίζοσπαστικοποίηση και την καταπολέμησή της. Ιδιαίτερα πρέπει να πούμε ότι έχουμε να κάνουμε με έκφραση και τοποθέτηση έναντι των νέων μέσω του διαδικτύου με μηνύματα μίσους. Αυτά πρέπει να καταπολεμήσουμε, βεβαίως με παρεμβάσεις ε, κοινωνικού ή και πολιτιστικού χαρακτήρα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μιλήσουμε και σε σχέση με την πιο τεχνική αυτή πλευρά που έχει να κάνει με την ε, απάλληψη ενδεχομένω των μηνυμάτων μίσου από το διαδίκτυο. Σε αυτό θα ήθελα την ε, δική σα αξιολόγηση για το κατά πόσον μπορεί να είναι σύμφωνη αυτή με την αντιμετώπιση και των θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα η αντιμετώπιση της προσωπικοποίησης στις φυλακές και γενικά τα σοφρονιστικά ιδρύματα έχει πολύ μεγάλη σημασία για μένα, το βλέπω και στη χώρα μου, σε θέματα και θρησκεία βεβαίω και κοινωνικά πρέπει να αντιμετωπιστεί η ροσπαστικοποίηση μέσα από τι φυλακέ. Και εκεί πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις για να αποφύγουμε την αντιστροφή μιας διαδικασίας η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο ομαλές εξελίξεις, ε, την αντιμετώπιση λοιπόν της ζωοπαστικοποίηση μέσα στα σοφινιστικά ιδρύματα. Θα ήθελα τις δικές σας απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ την Κατερίνα Κινίτση και παρακαλώ τον κύριο Φλάιρτη να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ε, μου είπε η πρόεδρος ότι θα παίξουμε πινκ-πονγκ με τις ερώτα απαντήσεις. Τώρα κατάλαβα τι εννοεί. Κυρία Κινίτση, σας ευχαριστούμε. Βεβαίως, η πράξη της ριζοσπαστικοποίησης είναι το θέμα σε πολλές περιπτώσεις, αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι πολύ ευρύτερο το πλαίσιο και αυτό είναι το τελευταίο στάδιο μόνο. Ε, δηλαδή δημιουργείται μια ευπάθεια στο άτομο και γι' αυτό αυτό το μήνυμα το διαδικτυακό ε, καταλαμβάνει και επηρεάζει το άτομο με τι εμπειρίες των μουσουλμάνων στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε, πρέπει να είναι ήδη κάποιοι αποξενωμένοι να νιώθουν ε, οργή, να μην νιώθουν ενταγμένοι στην κοινωνία για να ε, πιάσει αυτό το μήνυμα. Λοιπόν, εγώ για την αντιμετώπιση τη ρουσπαστικοποίηση θα πρότεινα να μην ασχολούμαστε με το τελευταίο στάδιο του μήνυματο, ε, γιατί αυτό σημαίνει ότι παραγνωρίζουμε ολόκληρα τα συμφραζόμενα, τα συγκείμενα, μια ιστορία που ξεκινάει από την παιδική ηλικία του ατόμου. Ε, αυτά για τη διαδικτυακή ριζοσπαστικοποίηση. Έχουμε την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, που υποστηρίζει ε, το να διαγράφονται από τις ιστοσελίδες τα μηνύματα μίσους. Εμείς, ε, ο δικός μας οργανισμός ε, ε, εξεργάζεται προγράμματα που φυσικά δεν κάνουμε εμείς η ίδια εκπαίδευση, αλλά φτιάχνουμε προγράμματα και modules τα οποία θα δώσουμε σε εθνικό επίπεδο για την για να μάθουν τα παιδιά ήδη στα σχολεία πώς να αναγνωρίζουν τις πλαστές ειδήσει για τον μεδιακό αλφαβητισμό. Ε, για τις ε, φυλακέ. ναι, ε, φυσικά δεν είναι αρμοδιότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δεν έχει σε αυτό το συγκεκριμένο τομέα παράξει έργο. Θα ήθελα μόνο να θυμίσω ότι υπάρχουν, υπάρχει και η παραγραφή, το θέμα της παραγραφή, όπως και για πολλές άλλες έξι πράξεις και όταν ή ε, μάλλον, συγγνώμη, το θέμα της νομιμοποίησης, ε, δηλαδή εάν ε, νομιμοποιείται ο στόχος που εσείς εντοπίζετε, τότε θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και να επεξεργαστούμε περαιτέρω το θέμα. Ευχαριστούμε κύριε Φλάερτη. Ο Ζεφρί Βανόρντεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Και, ε, Πρόεδρε, και ευχαριστώ κύριε Φλέρτη για τις παρατηρήσεις που κάνατε. Ε, είπατε να μην ε, εξισώνουμε, να μην συγχαίουμε τη μετανάστευση με την ασφάλεια. Συμφωνώ. Όμως για την Ισλαμική τρομοκρατία είναι αλληλένδετα αυτά τα δύο ζητήματα. Η πλειοψηφία των τρομοκρατικών πράξεων στο Ηνωμένο Βασίλειο την τελευταία δεκαετία διεπράχθησαν από ανθρώπους, ε, από μετανάστες ε, που έχουν, ε, ανθρώπους που έχουν μετικήσει στο Ενωμένο Βασίλειο. Αλλοδαπής προέλευση δηλαδή. Και βλέπουμε ότι παρόλα αυτά συνεχίζεται η μετανάστευση από χώρες που έχουν τελείως διαφορετική αντίληψη για το κράτος δικαίου και που ε, νιώθουν μια εχθρικότητα προς τις χώρες μας, έρχονται στις χώρες μας ε, και έχουν την εντύπωση ότι μπαίνουν σε κοινότητες ε, που τελικά ίσως και να είναι χειρότερες από αυτές που άφησαν και συνειδητοποιούν ότι αντί να ξεφύγουν από αυτό από το οποίο έτρεχαν τελικά παγιδεύονται από ομάδες εξτρεμιστών στην χώρα προορισμού, στη χώρα υποδοχής. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, θα πρέπει Πρώτα απ' όλα να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει αυτή η σχέση ανάμεσα στα δύο φαινόμενα και να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Ρωτώ, μήπως θα έπρεπε να επαναπροσδιορίσουμε κάποιες πτυχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το φως των προκλήσεων με τις οποίες ε, είμαστε αντιμέτωποι και ε, μιλώ και για υπαξιακής φύσης ε, προκλήσεις ενίοτε. Ε, απάντηση. Ευχαριστούμε κύριε Βανόρδεν. Δεν είμαι ε, σε θέση ε, να σχολιάσω συγκεκριμένα συμβάντα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν ισχύει ότι η πλειοψηφία αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών ε, έχουν διαπραγθεί από ανθρώπου πρώτη ή δεύτερη γενιά, δηλαδή αλλοδαπή προέλευση. Δεν ευσταθεί αυτό. και σε μεγάλο ποσοστό διαπράττονται από πολίτε των χωρών όπως σημαίνονται τρομοκρατική ενέργεια. Ε, και Ας μην ε, λοιπόν μετατρέπουμε σε πρόβλημα μια ολόκληρη κοινότητα ανθρώπων ε, όπως την κοινότητα των μεταναστών γιατί δεν έχουμε και εμπειρικά δεδομένα για να στηρίξουμε κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν ολόκληρη ομάδα να τύχει τη ίδια μεταχείριση επειδή κάποια μονομένα άτομα τη συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο. Ε, το 2015, παραδείγματο χάρη, που υπήρξαν μεγάλε πιέσει, σε 52% ε, έλαβαν διεθνή προστασία σε ε, επίπεδο πρωτοδικίου, πρωτού κατά κατατεθεί έφεση. Αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεφύγουν από ε, σειράξεις και χρειάζονται αυτή τη διεθνή προστασία. Ούτε όμως και ισχυριζόμαστε ότι σε αυτές τις κοινότητες δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Μα κακοί υπάρχουν και στις δικές μας, ε, ε, στη δική μας κοινότητα. Δεν το ισχυριζόμαστε αυτό. Όχι ότι δεν πρέπει να εξετάζουμε το θέμα της ασφάλειας, απλώς λέμε ότι δεν θα πρέπει να βάζουμε τίτλους. Δηλαδή, α, άμα είσαι μετανάστης, ε, είσαι και πρόβλημα και ε, τρομοκράτης. Ε, σε σχέση με αυτό που είπε ο κύριος Φανόρδαν, ότι είναι υπαρξιακές αυτές οι προκλήσεις, θα διαφωνήσω μαζί σας. Εγώ νομίζω πως θα πρέπει να δούμε σε ποιο βαθμό το διεθνές πλαίσιο μας προσφέρει η ευελιξία. Είναι ιδιαίτερα ευέλικτο ε, όργανο και στο διεθνές ε, ε, δημόσιο δίκαιο υπάρχει διαρκώς η ανάγκη εξισορρόπης των δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες και εμείς το μόνο που ζητάμε είναι να, υπάρχει, να ισχύουν οι αρχές της αλογικότητας, της νομιμότητας, της μη διάκρισης Μα το πινκ-πονγκ τι νόημα έχει. Θα πρέπει να μπορώ να επανέλθω και να δευτερολογήσω. Αλλιώ τι πινκ-πονγκ παίζουμε, λέει ο κύριο Φανόρδη. Ε, όχι, το πινκ-πονγκ ε, έχει την έννοια ότι όλοι οι συνάδελφοι έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν και ε, να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν. Η Άννα Γκόμες, ε, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, μα, ο όλος ο στόχος του εγχειρήματος είναι να μπορούμε να δευτερολογήσουμε. Αλλιώ δεν μπορούμε να το ονομάζουμε ping-pong. Θέλω να επανέλθω. Και δεν μου απάντησε ε, Εντάξει, το, αυτό, συμφωνώ με αυτό που είπε ότι και πολίτε των χωρών μα ε, ε, διαπράττουν αυτέ τι τρομοκρατικέ ενέργειε, αλλά θα πρέπει αυτή τη στιγμή να το αντιμετωπίσουμε το θέμα. Δεν δυσκολευόμαστε να ε, δεχτούμε ποιοι θα μπουν στη χώρα μα και ποιοι όχι. Και όταν ε, ε, τα, αναγνωριστούν ως εξτρεμιστές τους, θέλουμε να του απελάσουμε και μα εμποδίζουν οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό είναι το πρόβλημά μου, πρόεδρος. Ο κύριος Σοφλαέρτη απάντησε στην πρώτη σας ερώτηση. Συνεχίζεται η συζήτηση. Προτείνω λοιπόν να συνεχίσουμε για να μιλήσουν όλοι και για να λάβουν και τις απαντήσεις τους από τον προσκεκλημένο μας. Και αν στο χρόνο μας αναλογεί ε, περισσέψουν κάποια λεπτά, θα επανέλθουμε σε κάποια ζητήματα για να τα καλύψουμε όλα. Και αν δεν συμβεί αυτό ε, κατά διάρκεια αυτής της συνεδρίας θα το κάνουμε γραπτός. Ε, ο Γενικός Διευθυντή του οργανισμού ΦΡΑ έρχεται πάρα πολύ συχνά να μας δει. Ε, κυρία Γκόμες, ελπίζω να τηρήσετε το χρόνο σας αναλογή. Ε, thank Ευχαριστώ κύριε Φλέρτη που είπατε ότι χωρίς ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε αποτελεσματικά την τρομοκρατία γιατί τελικά και εμείς ε, πάμε στο ίδιο επίπεδο. Εγώ τουλάχιστον έτσι ερμήνευσα αυτό που είπατε. Και ευχαριστώ επίσης που τονίστε το θέμα της διάκρισης και της παρενόχλησης, γιατί πολλά από αυτά που αντιμετωπίζουμε ως προβλήματα στη δεύτερη και τρίτη γενιά έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτά. Και αυτά δυσκολεύουν την ένταξη των ε, μεταναστών στις κοινωνίες μας. Η ερώτησή μου είναι η εξής και έχει να κάνει με την ανάγκη ή διαφοροποίησης μέσα στις αστυνομικές δυνάμεις. Κυρίως όταν ακούμε από πολλούς που δουλεύουν με αυτά τα πράγματα που λένε ότι η, η ριζασπαστικοποίηση ουσιαστικά λειτουργεί ως εξής. Οι μεν τροφοδοτούν τους δε. Είναι ένας φαύλος κύκλος μουσουλμάνοι ή μετανάστες ανατροφοδοτούνται όσον αφορά την ριζοσπαστικοποίηση. Ποια είναι η άποψή σας από αυτού. Ευχαριστώ κυρία Κόμες για τα καλά σας λόγια επίσης. Πράγματι πρέπει να σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα στις στρατηγικές μας, όχι μόνο για να μην βρεθούμε και εμείς στο ίδιο επίπεδο με τους εγκληματίες, αλλά για να φροντίσουμε να έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την ασφάλεια. Έχουμε καλύτερη ασφάλεια αν δεν αποξενώνουμε τον κόσμο, αν δεν πλήττουμε την αξιοπρέπειά τους, αν δεν τους περιθωριοποιούμε. Συνεπώς, τα συστήματα ασφάλειας, αν ε, λειτουργούν ε, με σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δεν θα υπάρχει ζωσπαστικοποίηση. Έπειτα το θέμα της διαφοροποίηση μέσα στις αστυνομικές δυνάμεις, αν σας κατάλαβα καλά, αλλά και στο προσωπικό των φυλακών. Εντάξει, ναι. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι οι έρευνες μας δείχνουν όλο και περισσότερο ότι είναι πολύ σημαντικό οι κοινότητες αυτές να μπλέκονται. Και αυτό δεν γίνεται επαρκώς. Είναι πολύ δύσκολο και συγγνώμη αν επανέρχομαι στη δικιά μου εθνική εμπειρία, αλλά επειδή δούλεψα πάνω σε αυτά στη Βόρεια Ιρλανδία, διαπίστωσα ότι δεν φτάνει η καλή θέληση. Πρέπει να ξεπεράσει κανείς και ε, θέματα που έχουν να κάνουν με το ποιος κάνει τι στην κοινωνία και το χάσμα που υπάρχει μεταξύ γενεών πολλές φορές. Ευχαριστούμε πολύ για τις απαντήσεις σας, για τις εμπειρίες σας που μοιράζεστε μαζί μας. Ο Ζεράρ Ντεπρέτορα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Φλέρτη, δύο ερωτήσεις έχω για την διαλειτουργικότητα αναγνωρίσατε ότι μπορεί να είναι χρήσιμη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο οργανισμός σας δημοσίευσε μία έκθεση όταν δεν γνωρίζαμε ακόμα τις προτάσεις της Επιτροπής. Οι προτάσεις της Κομισιόν πια είναι γνωστές και προσπαθούν να ανταποκριθούν θετικά σε κάποιους κινδύνους που εσείς είχατε εντοπίσει και είχατε συστήσει στην Επιτροπή να εξετάσει. Τώρα τι θα κάνετε, την πρότασή σας θα την προσαρμόσετε, την ανάλυση σας πιο σωστά, βάσει της πρότασης που γνωρίζουμε πια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεύτερον, ο οργανισμός σας έχει κάτι να πει και για τη συζήτηση που γίνεται σε πολλές χώρες σήμερα για το κατά πόσο δηλαδή δεχόμαστε τους υπηκόους οι οποίοι έχουν πάει στη Συρία ή αλλού και έχουν συμμετάσχει εκεί στον πόλεμο. Πιστεύετε ότι εδώ υπάρχει θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να επιστρέψουν ή αντίθετα πρέπει να τους παραδώσουμε στη δικαιοσύνη στις διάφορες χώρες με ό,τι κινδύνους αυτό σημαίνει. Ευχαριστούμε. Παρακαλώ. Δύο ερωτήσεις κύριο Φλέρτη. Ευχαριστώ κύριε Ντεπρέ. Διαφορετικά σημεία. Πρώτον, για την διαλειτουργικότητα. Πράγματι, δώσαμε την ανάλυση μας στα πλαίσια των κλειστών εργασιών της ομάδας σε υψηλό επίπεδο. Κάποιες από τις προτάσεις μας, συστάσεις μας λήφθησαν υπόψη, κάποιες άλλες όχι. Κάποια στοιχεία στο κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν ε, είχαν ε, εξεταστεί στην ομάδα υψηλού επίπεδου. Όντως θα ήταν καλό ο οργανισμός μας να επανέλθει με παρατηρήσεις. Και έχουμε δύο δυνατότητες για να το κάνουμε αυτό. Η μία είναι του επόμενους μήνες να ετοιμάσουμε μια μεγάλη έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα βιομετρικά στοιχεία. Είναι κάτι που μπορεί να γίνει μέσα στους επόμενους δύο μήνες. Φυσικά πάντα είμαστε στη διάθεση του Κοινοβουλίου σας. Αν ε, θέλει την άποψή μας για ένα συγκεκριμένο θέμα, ευχαρίστως μπορεί και αυτό να γίνει, έτσι είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα για την επιστροφή των μαχητών, εγώ θα τους έλεγα ξένους μαχητές, γιατί ακριβώ δεν είναι ξένοι, είναι υπήκοοι χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό το εξετάζουμε στον οργανισμό μας. Η αρχική μου απάντηση εξακολουθεί να ισχύει ότι αν έχουν προβεί σε πράξεις, προφανώς και πρέπει να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Αλλά πρέπει να αποφύγουμε να καταλήξουν σε ένα καθεστώς απάτριδα. Είναι κάτι πάντως που εξετάζει ο οργανισμός μας αυτή την ε, εποχή. Ευχαριστούμε. Η Έλενα Βαλανθιάνο είναι η επόμενη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε, για τις εργασίες του οργανισμού σας και για οτιδήποτε συνεισφέρει τελικά προκειμένου η δικιά μας Επιτροπή να μπορέσει να εργαστεί σωστά. Γιατί το έργο μας δεν είναι απλό, ε. πρέπει και εμείς να καταλήξουμε σε προτάσεις που θα βελτιώσουν την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά που έχετε εσείς να μας πείτε. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα των χαμένων παιδιών μου έχει γίνει έμονη ιδέα μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση σύγχρονη, αναπτυγμένη, είναι απαράδεκτο να υπάρχει ένας ακαθόριστος αριθμός παιδιών που έχουν χαθεί. Γιατί αυτό λέμε, ότι έχουν χαθεί. Εντάξει, προφανώς δεν έχουν χαθεί. Έχουν πέσει στα χέρια μαφιόζων, λαθρεμπόρων κτλ. Θέλω να ξέρω λοιπόν περισσότερο για το τι κάνετε για αυτά τα παιδιά πώς συνεργάζεστε με την αστυνομία των χωρών μελών, τις ε, υπηρεσίες πληροφοριών των χωρών μελών κτλ. Γιατί από ό,τι φαίνεται είναι χιλιάδες αυτά τα παιδιά που έχουν χαθεί στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Βαλανθιάνο. Ναι, φυσικά και μας απασχολεί πάρα πολύ και μας το επίπεδο του αριθμού έτσι, των παιδιών αυτών. Αλλά έχουμε επίση την άποψη ότι μπορούμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά όσον αφορά την ιχνηλάτηση. Δηλαδή, πώ θα βρούμε τα ίχνη αυτών των παιδιών, διευκολύνοντα, για παράδειγμα, τι υποδομέ υποδοχή. Ακριβώ για να μην φεύγουν από εκεί τα παιδιά και χάνονται. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν διευκολύνσεις υποδοχής των παιδιών και καταλήμματος για τα παιδιά αυτά ε, πράγμα για το οποίο πρέπει να φροντίσουν άνθρωποι που έχουν ειδικευτεί σε αυτή τη δουλειά. Συνεπώ, πολλά μπορούν να γίνουν όσον αφορά την υποδοχή του και δεν έχει να κάνει με τη μία μόνο ή την άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κάνει με όλε. Γιατί από ό,τι φαίνεται, κάθε μήνα, στην ανάλυση που έχουμε κάνει, δηλαδή όσον αφορά τη μετανάστευση, βλέπουμε ότι παντού υπάρχουν τέτοια παιδιά. Δεύτερον, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχουν πολλά δεδομένα που μας επιτρέπουν να βρούμε τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε σε θέση να έχουμε μια διαδικασία για να βρούμε τα ίχνη αυτών των παιδιών. Είτε πρόκειται για τα δαχτυλικά αποτυπώματα στο Eurodac, είτε για κάποια άλλη βάση δεδομένων. Επειδή δεν έχουμε όμω τη διαλειτουργικότητα, δεν είμαστε σε θέση να εκμεταλλευτούμε και να συνδυάσουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Συνεπώ, η διαλειτουργικότητα, ο συνδυασμό δηλαδή όλων αυτών των πληροφοριών είναι ένα πολύ καλό νέο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα συστήματα κυδαιμονίας κατά κάποιο τρόπο για τα παιδιά αυτά πρέπει να λειτουργήσουν καλά. Δηλαδή τα παιδιά πρέπει να καλύπτονται και να μην εξαφανίζονται έτσι, να καλύπτονται από ένα τέτοιο σύστημα ε, αναδοχής ε, και ώστε ακριβώς να μην χάνονται αυτά τα παιδιά στη συνέχεια. Και υπάρχουν κάποιε βελτιώσεις σε πολλές χώρες μέλη τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα ο δρόμος που μένει είναι μακρύ, Δεν έχει διορθωθεί το πρόβλημα, αλλά βελτιώνεται, ακριβώς για να μην εξαφανίζονται άλλο τέτοια παιδιά. Α, και κάτι ακόμα για την ερώτηση της κυρίας Βαλανθιάνο. Ρωτάτε ε, τι κάνουμε για να βρούμε αυτά τα παιδιά. Ο οργανισμός μας, πρέπει να ξέρετε, δεν είναι λειτουργικός οργανισμός. Δηλαδή δεν έχουμε τη δυνατότητα, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε επί τόπου και να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα. Το λέω για να διευκρινίσω την κατάσταση, να το ξέρετε. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Στέφανης έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Φλάρτη για την παρουσία του εδώ σήμερα. Πράγματι πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι ζωτική σημασία να υπάρχει αυτή η ισορροπία. Και τώρα, κατά τα άλλα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, λέει ότι πρέπει να δίνονται τα δεδομένα. Και όντως οι υπηρεσίες πληροφοριών πρέπει να συνεργάζονται με την αστυνομία, κάτι το οποίο δύσκολα γίνεται σήμερα. Μιλάμε για θέματα ιδιωτικού βίου. Αν όμως αυτά τα δεδομένα δεν δίνονται στην αστυνομία, πώς θα δουλέψει η αστυνομία. Οπότε και εδώ πρέπει να υπάρχει καλή ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την προστασία του ιδιωτικού βίου και προσωπικών δεδομένων. Δεν λέω ότι πρέπει να ελευθερωθούν οι τρομοκράτες, αλλά όπως σας είπα και πριν, πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία. Ας πούμε ότι θέλει να εκδώσει μια χώρα έναν επίκο τρίτης χώρας, άλλης χώρας. Τι πρέπει να κάνουμε για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει σε μας. Γιατί είναι τα δικά του δικαιώματα πιο σημαντικά από τα δικαιώματα των θυμάτων. Αυτό θέλω να καταλάβω. Ευχαριστούμε. Ακούσατε έτσι τη μετάφραση, οπότε νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δύο θέματα θέσατε. Το ένα έχει να κάνει με την προστασία των δεδομένων και την προσέγγιση του δικαστηρίου και το δεύτερο έχει να κάνει με την προσέγγιση στους τρομοκράτες. Έτσι είναι δύο διαφορετικές ερωτήσεις, σωστά κατάλαβα. Οπότε θα επανέλθω και σε κάτι που ρώτησε νωρίτερο ο κύριος Φανόρδεν... που είχε την αίσθηση ότι δεν τον κάλυψα. Λοιπόν, πρώτα όσον αφορά τους κανόνες που διέπουν τα προσωπικά δεδομένα. Είναι αυτά που είναι. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει τοποθετηθεί, οπότε πρέπει να συμμορφωθούμε προς την απόφαση και να βρούμε τρόπους να κάνουμε την δουλειά μας προστατεύοντας την ασφάλεια, αλλά συμμορφούμενοι και προς την απόφαση του δικαστηρίου. Είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι το δικαστήριο δεν εμποδίζει το έργο των υπηρεσιών ασφάλειας. Το δικαστήριο αποφάσισε ότι η αρχική προστασία των δεδομένων δεν πρέπει να γίνεται αδιακρίτως, αλλά ότι μπορεί να γίνεται με αναλογικότητα και στοχευμένα βάσει διαφόρων παραμέτρων. Αυτό δηλαδή είναι ένα παράθυρο ανοιχτό για μας. Το άλλο είναι ότι η πρόσβαση στα δεδομένα αυτά μπορεί να επιτραπεί εφόσον δίνεται η άδεια βάση συγκεκριμένων προϋποθέσεων αφού προηγουμένως μια δικαστική αρχή είχε εξετάσει την υπόθεση και ανεξάρτητη υπουργική αρχή. Η απέτηση αυτή όμως αμβλύνεται εφόσον υπάρχει το κατεπήγον. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχει ένα παράθυρο ανοιχτό για μας. Τώρα, πέρα από την απόφαση του δικαστηρίου όμως για την προστασία των δεδομένων, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι υπάρχει και οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωση για την προστασία ε, των προσωπικών δεδομένων από τις αρχές συμμόρφωσης προς τον νόμο. Αυτό το οποίο θέλω να πω δηλαδή στους βουλευτές είναι ότι είτε πρόκειται για το τελεσβέρικα για άλλα συστήματα που έχουμε δεδομένων, δεν είναι όπως ακριβώς φαίνεται. Και για το θέμα της ε, έκδοσης. Υπάρχει η αρχή του non-refoulement, που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να διώξουμε ανθρώπους προς χώρες στις οποίες κινδυνεύουν από δίωξη εκεί. Αν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, δεν έχουμε το δικαίωμα να στείλουμε πίσω ανθρώπους. Η αρχή αυτή του non μία απόθεσης είναι μια από τις πιο παλιές αρχές. Είναι μια αρχή πολύ καλά ριζωμένη στα κράτη δικαίου που πρέπει να τηρούμε. Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας και τις διευκρινήσεις. Εν παρόδο για την πρώτη ερώτηση. Η κυρία Μπίρκετ Σίπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω ερώτηση για τη διαλειτουργικότητα γιατί δεν άκουσα πολύ σαφείς δηλώσεις σε σχέση με τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Συμφωνώ ως προς κάποιες από τις προκλήσεις που αναφέρατε, αλλά η εισαγωγή μόνο ευρωπαϊκής διαλειτουργικότητας για μένα δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Πρώτον λοιπόν, η ποιότητα των δεδομένων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Έχουμε ακόμα πολλά προβλήματα. Δεν είναι συγκρίσιμα τα δεδομένα, δεν είναι αναγνώσιμα από διαφορετικέ βάσει και αυτό είναι ένα κύριο πρόβλημα. Δεύτερον, δεν υπάρχει μια ενιαία γραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το πώ θα αποφασίζεται το ποια πληροφορία είναι τόσο σημαντική ώστε τελικά να πρέπει να μπει στο σύστημα ή ποια δεν είναι αρκετά σημαντική. Λέτε ότι θα πρέπει να επιληθούν κάποια προβλήματα, όντως. Αλλά ίσω να έχετε μάλιστα περισσότερε πληροφορίε ε, εσεί δεν και να μπορείτε να μου απαντήσετε. Αλλά πάντω εγώ δεν βλέπω πώ μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα αυτά. Και από την άλλη, η εξασφάλιση διαλειτουργικότητα προποθέτει κόστο, τεχνικέ τροποποίησει. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα πολύ συχνό, ότι δηλαδή είναι κακή η ποιότητα των δεδομένων, τόσο που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ή πολλέ φορέ καθυστερεί πολύ η εισαγωγή του εθνικέ βάσει δεδομένων. Ή αν εισαχθούν σε εθνικέ βάσει δεδομένων, δεν εισάγονται αντίστοιχα και στι ευρωπαϊκέ βάσει δεδομένων τα ίδια στοιχεία. Άρα λοιπόν πώς θα λυθεί το ζήτημα της διαλειτουργικότητας αν έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις. Δεν θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθούμε στην επίλυση αυτών των προβλημάτων και μετά να περάσουμε στο δεύτερο βήμα. Και αν καταφέρουμε όλα αυτά δεν θα έχουμε προχωρήσει σημαντικά, γιατί δεν πρέπει να κάνουμε το, το δεύτερο βήμα πριν από το πρώτο. Και Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε ακόμη μια-δύο προτάσεις για ένα άλλο διαφορετικό θέμα. Δεν υφίσταται αντιπαράθεση, πόλεμος μεταξύ θρησκειών. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Έχουμε πόλεμο μεταξύ ε, κέντρων εξουσίας. Οι δυτικέ χώρες ήταν εκείνες οι οποίες επηρέασαν χώρες με μουσουλμανική κουλτούρα και νοοτροπία και θέλω να υπενθυμίσω στους πάντες ότι το Ιράν είχε μπει σε ένα πολύ καλό δρόμο, αλλά στη συνέχεια οι Ηνωμένε Πολιτείε και το, Ευρωπαϊ... και το Ηνωμένο Βασίλειο παρενέβησαν στο Ιράν και έχουμε βρεθεί στην κατάσταση αυτή. Αντίστοιχες ε, συνθήκες έχουμε στο Αφγανιστάν, την ε, Συρία, στην Ιεμένη έχουμε μια αντιπαράθεση μεταξύ Πολιτείων και Ρωσίας. Δεν έχουμε να κάνουμε αντιπαράθεση με το μουσουλμανικό πληθυσμό. Επιπλέον, μεταξύ των προσφύγων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι έχουν πολύ καλά ε, έχουν χαρακτηριστικά που θα τους επέτρεπαν εύκολα να μπουν στο καθεστώς των προσφύγων, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από τις χώρες αυτές. Ας μην μπερδεύουμε λοιπόν διαφορετικά πράγματα και εδώ θέλω ιδιαίτερα να ε, υποστηρίξω τον κύριο Βλάερτη. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαιώματα και εγκληματίας ακόμη να είναι και τρομοκράτης να είναι, δεν επιτρέπεται να τον απελάβουμε, να τον στέλνουμε σε, μια χώρα που μπορεί να φωνευθεί. Πρέπει να τον πάμε στο δικαστήριο, ναι, να τον βάλουμε φυλακή, έχουμε δικαίωμα, ναι, αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε τα θεμελιώδη του δικαιώματα, λυπούμε πολύ. Αλλά πάλι επανέρχομαι, πρέπει να λύσουμε τα ζητήματα της διαλειτουργικότητας με τη σειρά πριν περάσουμε στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας. Η Πρόεδρος. Ευχαριστώ και σας δίνω το λόγο κύριο Φλαέρτη για τα ζητήματα αυτά που έχουν και τεχνικό χαρακτήρα. Και βέβαια οφείλονται σε ένα μεγάλο βαθμό και στη γενικότερη κατάσταση και τι συνέπειέ τη στην τρομοκρατία. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Ζήπη για τις ερωτήσεις για τη λειτουργικότητα ε, στα σχόλιά μα τα γραπτά που έχουμε ήδη δημοσιεύσει που σχετίζονται βέβαια με τις προτάσεις που διατυπώσαμε και συζητήσαμε κατά το καλοκαίρι και από αυτά που τα οποία έγιναν δεκτά τώρα από την Επιτροπή έχουμε να κάνουμε μια διευκρίνηση ε, με τα μεταγενέστερη. Έτσι λοιπόν μπορεί να υπάρχουν κάποια θέματα στα οποία δεν έχουμε τοποθετηθεί. Αλλά πάντως στην ε, λεπτομερή μας ανάλυση, της οποίας μόνο μια γενική γεύση σας έδωσα σήμερα, αλλά βέβαια είναι διαθέσιμη, είναι δημοσιευμένη ε, στη διάθεση των βουλευτών, επισημαίνουμε την αναγκαιότητα και την αναλογικότητα ω βασικές αρχές και εδώ ακριβώς ε, έρχεται το σύστημα της ε, αλληλουχίας που προτείνουμε ως προς την ε, διαλειτουργικότητα, δηλαδή τα διάφορα στάδια για να εξασφαλιστεί αυτή και μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση που πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί, που ανάφερα και νωρίτερα, που έχει να κάνει με τον περιορισμό ως προς τον σκοπό των μέτρων. Επίσης, η ποιότητα των δεδομένων μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί ιδιαίτερα. Το ανέφερα και νωρίτερα πως υπάρχουν στοιχεία ότι φύστανται σφάλματα. Το ότι διαπράττονται σφάλματα σημαίνει όχι μόνο καταστροφικές συνέπειες για τις ανθρώπινες ζωές, αλλά και ε, ε, αποδυνάμωση των συνθηκών ασφαλεια για την ίδια την Ευρώπη. Στην έκθεση βιομετρικών δεδομένων, παραδείγματι, θα σας παραπέμψω για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτηματικά των βουλευτών. Ευχαριστώ πολύ, Μπέρν Κιόλμελ, για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ και εγώ τον ε, κύριο Ιφιντή. Νομίζω ότι δεν διαφωνεί κανείς στη διαπίστωση ότι κάθε άνθρωπος έχει αναπαλωτρίωτα ανθρώπινα δικαιώματα ανεξαρτήτως ε, της όποιας υπετιότητάς του σε αδικήματα. Ταυτόχρονα όμως θέλω να επανέλθω στα όσα είπε ο κύριος Φανόρτεν νωρίτερα ότι ιδιαίτερα στον τομέα της ε, τρομοκρατίας και παρακαλούμε με παρεξηγήσετε δεν μπορούμε να έχουμε μόνο μια θεωρητική προσέγγιση. Πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε με τι πολύ συγκεκριμένα προβλήματα έχουμε να κάνουμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη χρονική στιγμή. Και εδώ βεβαίως έχουμε να κάνουμε με τον τομέα της μετανάστευσης που αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του φαινομένου της τρομοκρατίας χωρίς αυτό να σημαίνει ότι συμψηφίζουμε ή ότι ε, ταυτίζουμε την τρομοκρατία με τη μετανάστευση, ότι η μετανάστευση οδηγεί σε τρομοκρατία, η τρομοκρατία σε μετανάστευση. Α, μπορεί να μην ισχύει αυτό, αλλά η τρομοκρατία οπωσδήποτε επηρεάζεται από τα, τα μεγάλα νούμερα των μεταναστών που έρχονται, που έχουν έρθει και που θα συνεχίσουν να καταφθάνουν στις χώρες μας. Έτσι λοιπόν, οπωσδήποτε είναι πολύ σωστό το ότι χρειάζεται μια καλή ένταξη στις κοινωνίες ε, και αυτή αποτελεί το καλύτερο μέτρο κατά της τρομοκρατίας. Ταυτόχρονα όμως, και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό γιατί θέλω να το ακούσω από το στόμα σας, ότι υπάρχουν κάποια όρια του εφικτού, δηλαδή δεν μας εξυπηρετεί σε τίποτα και θα απογοητευτούν πολλοί οι πολίτες μας και ψηφοφόροι, εάν τους, μετα... αν τους περιγράψουμε ένα μόνο θεωρητικό ε, μοντέλο, στο οποίο όμω βλέπουν ότι όσο καλό και να είναι, δεν είναι υλοποιήσιμο και ρεαλιστικό. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ποια είναι τα όρια του εφικτού και αν έχουμε την εντύπωση, αν έχει ο πολίτης ότι έχει την εντύπωση ότι δεν είναι εφικτό να ξεπεράσουμε κάποια συγκεκριμένα θεωρητικά όρια, τότε ίσω θα πρέπει, ίσως ενδεχομένω, θα πρέπει σε κάποιο σημείο να υπάρχουν τροποποιήσεις και προσαρμογές στο νομοθετικό πλαίσιο. Εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε θέση να καταφύγουμε σε κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Και θα ήθελα από εσά να ακούσω ε, μια περιγραφή των τομέων, των ε, σημείων στα οποία μπορείτε να έχετε μια καλύτερη, μπορείτε να προσφέρετε ή να δείτε καλύτερη ανταλλαγή ε, δεδομένων και για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας και γενικότερα της εγκληματικότητας και βεβαίως αυτό θα πρέπει να αξιοποιηθεί ε, ασφαλώς όχι μόνο για την αντιμετώπιση τρομοκρατίας στο πλαίσιο της μετανάστευσης αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στον πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο στον τομέα αυτών. Χρειάζονται λοιπόν σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένα μέτρα τα οποία να είναι και υλοποιήσιμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει, πρόεδρος και ειδού μια πυκνή ερώτηση, φαντάζομαι και η απάντηση από πλευρά σας θα είναι αντίστοιχη. Κύριο Σουφλάρτη, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όντω, ευρύτατο το φάσμα των ζητημάτων που καλύψατε. Στα θέματα τη προστασία των δεδομένων και ε, διακράτησης δεδομένων, παρέπεμψα ήδη στι ε, πολύ λεπτομέρειε κατευθυντήριε γραμμέ που μας έχει ήδη εκδώσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αλλά και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων που προσφέρουν ε, ύψιστε υπηρεσίε στον τομέα και στην καθοδήγηση για το τι θα πρέπει να γίνει και για να υπενθυμίσω ακόμη το ότι δεν έχει αποκλείσει πρόσβαση σε δεδομένα το δικαστήριο, αλλά έχει δώσει ένα κατάλογο ε, μέτρων με βάση τα οποία μπορούν, μπορεί να εξασφαλιστεί θεμητή και νομίμη πρόσβαση στα στοιχεία. Ως προς την κοινωνική ένταξη. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως ε, την ερώτηση του κ. Κέλνερ και σε σχέση με, την, ε, με, το θεμελιώδη χαρακτήρα και τη θεμελιώδη σημασία της κοινωνικής ένταξης. Υπάρχουν βέβαια κάποια κέρια ζητήματα που αναδύονται διαρκώς, παραδείγματι ε, η de facto, ο de facto διαχωρισμός, ο κοινωνικός διαχωρισμός και αποκλεισμός και στη στέγη αλλά και στην εκπαίδευση. Ένα ιδιαίτερο παράδειγμα θα είναι αυτό τον Ρωμά. Μπορεί να μην γίνεται εσκεμένα, αλλά γίνεται de facto ε, και επειδή δεν έχουμε επαρκεί σπόρους για την ε, γλωσσική εκπαίδευση των νέων αφιχθέντων μεταναστών. Ένα μετανάστη που έρχεται σε μια χώρα και δεν γνωρίζει τη γλώσσα τη, δεν έχει το περιθώριο να πληρώσει μαθήματα γλώσσα ακριβά πολλέ φορέ για να ε, μάθει την ε, νέα αυτή ε, γλώσσα και βέβαια δεν έχει δυνατότητες για ένταξη στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε ταυτόχρονα και ο κύριος Γκόλνερ αναφέρθηκε σε μια θεωρητική προσέγγιση. Ναι, είναι θεωρητική η προσέγγιση, συμφωνώ, χρειάζεται μια πιο εφαρμοσμένη προσέγγιση στη δουλειά μας, τι φέρνει αποτελέσματα και τι όχι. Και σε αυτό ακριβώς αναφερόμαστε σε ε, προσπάθειες σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο πόλεως, όχι σε επίπεδο πρωτεύουσα κεντρικό. Πρέπει οι τοπικές κοινωνίε να ε, κάτσουν να συζητήσουν με τους εκπροσώπους ε, και τα μέλη της κοινωνίας των μεταναστών για να δουν ποιε είναι οι πιο αποτελεσματικές λύσεις. Ένα από τα σημαντικά έργα λοιπόν της υπηρεσίας μας και της ε, δουλειά που κάνουμε μέσα από τις εκθέσεις μας είναι να καταγράφουμε τις πλέον υποσχόμενες μεθόδους συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο στα διάφορα κράτη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ε, κύριε Διευθυντά. Για να ολοκληρώσουμε αυτό τον πρώτο γύρο και θα σας ξαναδώσω το λόγο στο δεύτερο γύρο για όσους θέλουν να θέσουν ερωτήματα ping-pong. Όχι ότι θέλουμε να σας, σας ένα μαρτύριο για σας απλώς είναι ένα σύστημα που έχουμε εφεύρει ε, για να ε, έχουν τη δυνατότητα ε, με βέλικτο τρόπο να θέτουν τα ερωτήματά τους οι συνάδελφοι. Ο κύριος Φροντσουλικά. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε Διευθυντά για την ε, παρουσίασή σας. Ε, αποσκοπούμε στην οικοδόμηση μιας ένωσης ε, της ασφάλειας ε, σε συνεργασία όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι άγνωστο προς το παρόν ποια μορφή θα λάβει αυτή η ένωση, ο χώρος ασφάλειας. Αυτό που πάντως επιθυμούμε είναι να αναβαθμίσουμε την ασφάλεια των πολιτών λαμβάνοντας υπόψη τις παρελθούσες ε, προκλήσεις και προβλήματα. Κυρίως ε, μετά την έκθεση ε, του Κοινοβουλίου το 2014 με τις μαζικές παρακολουθήσεις και την έκθεση που εξέδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, είχατε αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα σε σχέση με αυτό και δώσατε συγκεκριμένε απαντήσεις εκείνη την εποχή. Και θέλω να σας ρωτήσω ε, ανάμεσα σε αυτές τις μαζικές παρακολουθήσεις ε, με τα μέσα επικοινωνιών, κάτι που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε απειλές, κυρίως την απειλή της τρομοκρατίας, και από την άλλη πλευρά της πλάστικας έχουμε την ε, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών και των μεταναστών μεταξύ αυτών. Ε, πώς θα βρούμε την ισορροπία, δεν χρειάζεται μία νομοθεσία, ένα νομοθέτημα ή τουλάχιστον κάποιους ε, κοινού κανόνες για τα συστήματα παρακολούθησης και υποκλοπών, διότι κάποιες χώρες έχουν τέτοιους κανόνες, άλλες όχι και είναι δύσκολο να ε, παραβλέψουμε τις θέσεις των κρατών για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστούμε. Απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ο οργανισμός, κατόπιν ετήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έξω μία έκθεση για ε, το θέμα ακριβώς αυτό. Παρακολουθήσει στα κράτη-μέλη. Ε, είναι μία, δύο, τόμοι, δύο τόμους αριθμοί αυτή η έκθεση πριν από κάποια χρόνια ο πρώτος και μετά πάλι ε, εκδόθηκε και ο δεύτερος τόμος μετά από αίτημα του Κοινοβουλίου. Και υπάρχουν κάποια θέματα που ε, με όχι μεγάλη δυσκολία θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο κρατών μελών. Παραδείγματο χάρη, ε, υπάρχουν νομοθεσίες για στοχευμένες παρακολουθήσεις, ε, αλλά για τις, τις, αφ, τις μη ε, προγραμματισμένες παρακολουθήσεις δεν τις καλύπτουν αυτά τα νομοσχέδια και φυσικά πρέπει να ισχύει η αναλογικότητα, η ισότητα, η μη διάκριση αλλά ε, πρέπει να ισχύει και η νομιμότητα και αυτό δεν ε, κατοχυρώνεται αν δεν υπάρχει καν νομοσχέδιο που να καλύπτει κάτι όπως αυτό των μη προγραμματισμένων υποκλόπων οι αρχέ εποπτείας των κρατών μελών. Νομίζω υπάρχουν πολύ καλές πρακτικές στα κράτη-μέλη ως προς τις δεξιότητες, τα, ε, τους ε, την πρόσβαση και μπορούμε να μάθουμε πολλά από άλλα κράτη-μέλη. Και επίσης ε, τα ένδικτα... Ε, η τιμωρία και τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όταν είναι παράνομη η παρακολούθηση και η υποκλοπή. Ε, αυτό είναι στον αντίποδο του δεύτερου ζητήματος ε, και ο οργανισμός δεν θα συνεχίσει να επεξεργάζεται αυτό το ζήτημα. Απλώς σας ανέφερα τώρα κάποια ζητήματα που εμπειρεύονται σε αυτούς τους δύο τόμους της έκθεσης που εκδώσαμε. Σας ευχαριστούμε. Θα ήθελα κι εγώ να επανέλθω και να σας θέσω μία ερώτηση που όχι ότι θα ήθελα να ε, θίξω κάποιο ευαίσθητο θέμα, απλώς ε, για τη διαλειτουργικότητα, επειδή το έθιξαν οι συναδελφοί ε, άμεσα ή έμεσα και είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, είναι στην μέση διάταξη του Κοινοβουλίου, απηχώντας και το έργο του οργανισμού σας. με μεθοδικό, σχεδόν παιδαγωγικό τρόπο θα ήθελα να σας ρωτήσω και διευθυντά ποια ε, είναι τα στοιχεία που έχετε ήδη ε, αξιολογήσει ε, θα μας βοηθούσε πολύ για να βρούμε μια ισορροπία και να δούμε πού υπάρχουν ατέλειες στα συστήματά μας να έχουμε κάποια, την άποψη των, του, του οργανισμού, την ε, πραγματογνωμοσύνη του οργανισμού. Εφόσον μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να ε, διαβουλευτούμε και αν δεν μπορείτε ε, σήμερα, μπορείτε ε, να μας στείλετε στοιχεία διότι η πρόταση επιτάπητος ε, καλύπτει τα ζητήματα που ήγηραν οι συνάδελφοι ε, στα ερωτήματά σας. Δεν, μου είχαν βάλει το χρονόμετρο, δεν νομίζω να ξεπέρασα το ένα λεπτό. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μιλαντσφέ. Αν έχετε την καλοσύνη, θα ήθελα να απαντήσετε στο ερώτημά μου, κύριε Συντά. Ευχαριστώ. Εμείς ε, είδαμε μόνο ε, το Δεκέμβρη στο τέλος ε, την πρόταση επιτροπής και έχουμε κάνει μια περιορισμένη και προκατακτική ανάλυση μόνο. Παρ' όλα αυτά ήδη εντοπίσαμε δύο ζητήματα όπου θα πρέπει να δείξουμε εγρήγορση, ας το θέσω έτσι. Δύο στοιχεία που προτείνονται τώρα που ε, δεν έχουν αναλυθεί από την ε, ομάδα υψηλού επίπεδου. Υπάρχουν ίσω και περισσότερα, αλλά εγώ ε, δύο υπέπεσαν στην αντιλήψή μου. Ο ανοιχνευτή πολλαπλών ταυτοτήτων και ο εντοπισμός επικών τρίτων χωρών για λόγους δημόσιας ασφάλειας όπως αυτό ορίζεται στην Εθνική Νομοθεσία τα δύο θέματα θα πρέπει να τα προκολουθήσουμε εκ του να είμαστε δηλαδή σε ε, ε, εγρήγορση, γιατί δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, δεν μπορεί να υπάρξει έλεγχος. Ε, σε κάποια σημεία λύθηκαν υπόψη οι προτάσεις μας, σε άλλα όχι. Θα σχολίαζα το θέμα αυτό που αναφέρατε και εσείς για τα λάθη και την τιμωρία, διορθωτικά μέτρα. Ε, θεωρούμε ότι στο έγγραφο της Επιτροπής θα μπορούσε να ε, αποδοθεί μεγαλύτερο βάρος αυτό. Κυρίως, ε, κυρίως στην περίπτωση, σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται παιδιά. Διακράτηση δεδομένων για τα παιδιά. Ισχύουν διατάξει που δεν ισχύουν για του ενήλικε. Παραδείγματο χάρη, με παράνομη διέλευση των συνόρων υπό την εποπτεία ενό γονιού. Αυτό το παιδί, γιατί να ε, ε, νέο είναι έξι μηνών, γιατί να το έχει στο φάκελό του αυτό για ολόκληρο, τη ζωή. Ε, θα πρέπει να διαγράφονται αυτά τα δεδομένα κάποια στιγμή. αυτή είναι η προκατακτική ανάλυση, δηλαδή ότι μπορούμε να εντοπίσουμε τέτοιες ανησυχίες και να τις διορθώσουμε στο έγγραφο, στην πρόταση της Επιτροπής. Επίσης, προτείνουμε υπάρχει μεγαλύτερο σεβασμός ε, για την αρχή της ε, Αναλογικότητα. Ε, θέλουμε στο πλαίσιο της διαλειτουργικότητας να υπάρχουν διάφορα στάδια. Ε, δηλαδή, γιατί ο σύστημα Eurodac, παραδείγματος χάρη, ε, μόνο, ε, θα κατοχυρωθεί ότι δεν, μπορεί να, ε, δεν, δεν ε, υπάρχουν τα δεδομένα σε βάση δεδομένων που χρησιμοποιούνται από τις αρχές επιβολής νόμου και μόνο τότε θα υπάρχει πρόσβαση στη Eurodac. αυτό, γι' αυτό μιλάμε για το cascade, δηλαδή για την σταδιακή πρόσβαση, χορήγηση πρόσβασης στα, στις βάσεις δεδομένων. Ε, και εν ευθέτω χρόνο θα επανέλθω και σε κάποια από αυτά τα ζητήματα. Σας ευχαριστώ που με διαφωτίσατε κύριε Διευθυντά για αυτό το ζήτημα. Το σημειώνουμε ε, και πιστεύω ότι θα μας δοθεί και πάλι ευκαιρία να συζητήσουμε για την εξέβρεση αυτής της ισορροπίας, γιατί είναι εργαλεία που όντως χρειαζόμαστε για την καταμολέμηση της τρομοκρατίας, κυρίως αυτό το θέμα που ε, θίξατε για τις πολλαπλές ε, ταυτότητες στη Γαλλία, στη χώρα μου, στη τελευταία τρομοκρατική ενέργεια. Ε, διαπιστώσαμε όλοι πόσο εύκολο είναι να έχει κάποιος πολλές ταυτότητες και όντως θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, αξιολόγηση για να μπορέσουμε ε, αποτελεσματικά να προστατεύσουμε τους πολίτες από αυτό το φαινόμενο. Μίλαν Σφέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση της έρευνάς σας. Με παρακολουθείτε? Ωραία, ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι έχω μία ερώτηση. Γνωρίζω το έργο σας, γνωρίζω το έργο του οργανισμού σας στην Βιέννη. Έχουν γίνει πολλά τα τελευταία χρόνια για την προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων. Όμως, θα ήθελα να μοιραστώ μια σκέψη μου μαζί σας. Κάτι που μου απασχολεί, να πάση περιπτώσει, εδώ και καιρό. Ο οργανισμός σας θα έπρεπε ή ασχολείται τέλο πάντων με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ωραία. Όταν όμως διαβάζουμε τις εκθέσεις σας, διαπιστώνουμε συχνά ότι αντί να ασχολείστε με τα θεμελιώδη δικαιώματα, συχνά ασχολείστε με τα δικαιώματα των ανθρώπων δεύτερης και τρίτης γενιάς. Πολιτιστικά δικαιώματα, δικαιώματα πολιτιστικών ε, μειονοτήτων, ε, ατόμων ΛΟΑΔΑ, ομοφιλόφιλων δηλαδή κλπ. Οπότε διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλά θέματα που δεν έχουν διευθετηθεί μέχρι τώρα. Θέματα ιδιοκτησίας, για παράδειγμα. Μετά από 25 χρόνια, υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων που το 1945 έγινε κατάσχεση ε, περιουσίας, αλλά δεν έχει αποδοθεί ακόμα. Ή θέματα άλλα δικαιωμάτων. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα προτιμούσα εσείς να ασχολείστε και με τέτοια θέματα ε, προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Διευθυντής για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να διευκρινίσω πώς επιλέγει τα θέματα του ο Φυσικά πάντα προσπαθεί να προστατεύσει τους ανθρώπους που είναι περισσότερο ε, περιθωροποιημένοι, αλλά πρωτίστως ενδιαφέρεται για την προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων διαφόρων κοινοτήτων. Δηλαδή φυσικά και θέλουμε να υποστηρίζουμε και να προστατεύουμε τα δικαιώματα των πιο περιθωριοποιημένων ανθρώπων, αλλά τότε ξέρουμε ότι πρόκειται για τους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εμείς ασχολούμαστε και με ε, κοινότητες που έχουν πιο γενικά δικαιώματα προς προστασία των αναπήρων, για παράδειγμα. Ο Μιλοάδ είναι μια άλλη περίπτωση. Γι' αυτό και ασχολούμαστε και όλο και περισσότερο με τα κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα στα πλαίσια του κοινωνικού πυλώνα. Βέβαια, περιοριζόμαστε σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε, επειδή υπάρχουν περιορισμοί στον κανονισμό μας. Για παράδειγμα, το πολιετές πλαίσιο που θέτει περιορισμούς για τα θέματα τα οποία μπορούν να μας απασχολήσουν. Και εμείς τις δραστηριότητε μας τις εντάσσουμε σε αυτά τα πλαίσια. Αν το θεματικό δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο αυτό, ε, δεν μπορούμε να ασχοληθούμε με αυτό. Επίσης, κάτι άλλο που μας περιορίζει στις δραστηριότητε μας είναι το γεγονός του, το ότι υπάρχει ο τρίτος πυλώνας. Δηλαδή, δεν μπορούμε η Δία Πρωτοβουλία να αναλάβουμε έργο ε, στο τομέα της αστυνομίας. Και εκεί εμπίπτει και το θέμα ε, της δίκαιας δίκης Πολύ θα θέλαμε να μην υπάρχουν αυτοί οι περιορισμοί και μακάρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μας στηρίξει στο αίτημα μας αυτό για να μπορούμε να ασχοληθούμε με πολύ περισσότερα θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που απασχολούν τις κοινωνίες μας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Διευθύντα και για την απάντηση και για ε, τους ε, δρόμους που μας προτείνετε για να προχωρήσουμε. Τέλος, θα δώσω το λόγο στον κύριο Βανόρντεν επειδή ζήτησε να ξαναπάρει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριο Φλάρτη, επιβεβαιώνεται ότι ρόλο σας είναι να προστατεύετε τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Πιστεύω εγώ ότι η προτεραιότητά μας θα πρέπει να είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα ολόκληρου του πληθυσμού. Η συζήτησή μας, οι απαντήσεις που πήραμε έχουν να κάνουν με την τρέχουσα νομοθεσία και την ερμηνεία που δίνεται σε αυτή. Το έργο της δικιάς μας Επιτροπής είναι να προτείνει αλλαγές που θα πρέπει να γίνουν. Αλλιώς τι νόημα έχει να έχουμε μια τέτοια Επιτροπή. Οπότε, εσείς αναγνωρίζετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιας αλλαγής, προσαρμογής της νομοθεσίας που έχει να κάνει με την προστασία των δικαιωμάτων υπό το φως της τρομοκρατίας. Ο κύριος Σοφλάρτη. Ευχαριστώ. Με κάθε σεβασμό, αλλά δεν είναι ότι θέλω να πω κάτι αυτή τη φορά, έτσι. Αναρωτιέμαι αν με ακούτε κύριε Βανόρδεν, γιατί νομίζω ότι το ρητά ότι εμείς εξυπηρετούμε τα θεμελιώδη και ανθρώπινα δικαιώματα κάθε δικαιοδοσίας ε, στην οποία εμπίπτει το έργο μας. Απάντησα για το ότι αυτό πρέπει να φανεί ακόμα περισσότερο λαμβάνοντα υπόψη το καθήκον μας να προστατεύουμε τα δικαιώματα του συνολικού πληθυσμού. Εμείς βέβαια προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πιο ευάλωτους, αυτούς που βρίσκονται περισσότερο στο περιθώριο. Αυτή είναι η προτεραιότητα που δίνουμε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με τους Ρώμα, γι' αυτό ασχολούμαστε με τα παιδιά που έχουν χαθεί, όπως λέμε. Ε, θέματα δηλαδή τα οποία αποτελούν προτεραιότητα ακριβώ επειδή είναι πιο ευαίσθητα. Δεν είναι ρόλος του οργανισμού μας να αποφασίζει θα σας πω την προσωπική μου άποψη. Υπό το Βασίλειο προσπαθήσαμε να θέσουμε τα πλαίσια για τα οποία μπορεί να είναι περήφανη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα, πώς λειτουργούμε και τι αποτελέσματα φέρνουμε. Και νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι για αυτά. Και πρέπει εδώ να μιλήσω και για τον Winston Churchill και για πολλούς άλλους πολιτικούς που μας βοήθησαν θέτοντας τα πλαίσια να φτάσουμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Αυτή είναι μια απάντηση που παρακάμπτει την ουσία θα έλεγα. Νομίζω ότι εδώ πέρα θίξαμε πάρα πολλά θέματα. Σας ευχαριστώ όλους και κυρίως εσάς που ήσασταν στη διάθεσή μας να έρθετε εδώ και να μιλήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν για το χρόνο που μας διαθέσατε και ευχαριστούμε που δεχτήκατε και αυτό το σύστημα ping-pong που λέμε ότι είναι ένα αθλητικό σύστημα αλλά είναι κάτι παραπάνω από αυτό. Και είναι νομίζω πολύ ευχάριστο για τους συναδέρφους, γιατί έτσι έχουμε ζωντανό διάλογο. Ευχαριστούμε πολύ λοιπόν. Και θα περάσουμε σε λίγο στον κύριο Τουιμπό που έχει ήδη φτάσει. Eh Σας ε, ευχαριστώ με μεγάλη χαρά. Υποδεχόμαστε τον υπερασπιστή των δικαιωμάτων, όπως είναι ο τίτλος του Ζακ Τουμπον, αγαπητέ Ζακ, αγαπητοί συνάδελφοι, για το δεύτερο αυτό τμήμα της συνεδρίασης της Επιτροπής μας. Βασπασίρτ, τι συμβαίνει. Μην Βασερ θέλετε. Α, Σπρίτσβάσερ θέλετε, ανθρακούχο νερό. Καλώς ορίζουμε λοιπόν τον Ζακ ε, Τουμπού, υπερασπιστών δικαιωμάτων στη Γαλλία. Και εξ ονόματος όλων μας σας ευχαριστώ που ήρθατε να μας μιλήσατε στις αρχές του 2018 στη συνεδρίασή μας. είσαστε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, αν όχι κάθε μέρα, πάντως πολύ συχνά στη Γαλλία. Και ο Ζακ Τουμπό είναι βέβαια πολύ γνωστή πολιτική προσωπικότητα, παρά την ε, μετριοφροσύνη του εγώ θα το πω και θα το υπενθυμίσω. Έχει σταδιοδρομία και κοινοβουλευτική, αλλά και σε κυβερνητικούς θόκους πρώτης τάξης σταδιοδρομία. Αγαπητέ Ζακ, πολλές φορές υπηρετήσατε και στη έδρανα της Εθνοσυνέλευσης της Γαλλικής και στα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή στις πολυθρόνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μεταξύ 2004-2009. Πολλοί συνάδελφοι σας θυμούνται και έχουν συνεργαστεί μαζί σας και βεβαίως εν τέλει ε, καταλαμβάνει και τις ιδιαίτερα σημαντικές αυτές υπηρεσίες του Υπουργείου του Πολιτισμού και της Γαλλοφωνίας στη Γαλλία. Θα θυμάστε φαντάζομαι τους αγώνες που έκανε για την πρόσπιση της γαλλικής γλώσσας και της ε, ε, διατύπωσης all good όπως ονομάστηκε. Συνεχίζει λοιπόν να αγωνίζεται για την πολυγλωσσία μεταξύ του 2013 και του 2015. Ήταν και υπουργό Δικαιοσύνης ταυτόχρονα από το 2015 έως το 2017 ο Ζακ Σε σχέση λοιπόν με τα θέματα της δικής μας Επιτροπής, είναι ιδιαίτερα ενήμερος. Το 2014 από τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας προτάθηκε η υποψηφιότητά του για τα καθήκοντα του υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ε, Εθνοσυνέλευση, που ενέκρινε, Εθνοσυνέλευση και Γερουσία μαζί, αυτή την εντολή, την εξαετή για τον Ζακ και έτσι ανέλαβε καθήκοντα τον Ιούνιο του 2014. Άρα είσαστε περίπου στο ίμιση της θητής σας, έχετε ήδη εκτίσει 3,5 χρόνια της εκτίας σας ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων. Δικαιωμάτων των πολιτών έναντι της διοίκησης, αλλά ταυτόχρονα και δυνάμει του νόμου έχετε στη θέση σας ιδιαίτερα σε εξουσίες ως προς την προαγωγή των δικαιωμάτων, δικαιωμάτων του παιδιού, που αναφέρθηκαν ε, ως προτεραιότητες, ιδιαίτερα ε, καταπολέμηση των διακρίσεων, σεβασμό της δεοντολογίας και αυτό που μας ενδιαφέρει πρωταρχικά σήμερα, ιδιαίτερες εξουσίες και δραστηριότητες σε θέματα ασφάλειας και άνθρωπινων δικαιωμάτων. Το νομοθετικό διάταγμα στο οποίο στηρίζεται η πολιτική για την καταπολέμηση τρομοκρατίας στη Γαλλία ε, δίνει στο Ζακ Τουμπον την ευκαιρία και να αποδείξει και να επιδείξει πόσο πλήρης ε, είναι η δραστηριότητα και ποικίλη η δραστηριότητα και η προσωπικότητά του, αλλά ταυτόχρονα και να επιδείξει την μεγάλη αμεροληψία και επαγρύπνηση του για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών εναντίασδήποτε ε, παραβίασης και κατάχρηση εις βάρος των δικαιωμάτων του και κυρίως σε σχέση με την ανάλυση των τεχνολογιών, της τεχνικής, των υπηρεσιών πληροφορίας, πληροφοριών αλλά και της χρήσης του καθεστώτος της ανάγκης σε σχέση με τους περιορισμούς στην κυκλοφορία, την, ε, τον κατοίκο εγκλισμό και άλλα ζητήματα σε σχέση με την τρομοκρατία που είναι ιδιαίτερα επίκαιρα, ιδιαίτερα βέβαια στη Γαλλία αλλά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με μεγάλη χαρά λοιπόν σας υποδεχόμαστε εδώ, Ζακ Τουμπό. Μπορείτε να μας διαφωτίσετε σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της τρομοκρατίας που απασχολεί ιδιαίτερα την Επιτροπή μας, την ειδική αυτή Επιτροπή. Και με μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε την παρουσίαση και την προσέγγιση που θα μας ε, παρουσιάσετε. Και βέβαια ελπίζουμε ότι δέχεστε και εσείς αυτή την τεχνολογική του ping-pong που είδατε πώς λειτουργεί. Εάν τη δεχτείτε ασφαλώς θα μας διευκολύνει ιδιαίτερα στις εργασίες μας και θα εμπλουτίνει τη συστήση μας σήμερα. Σας δίνω λοιπόν αμέσως το λόγο κύριε υπερασπιστά των δικαιωμάτων. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ξεκινώντας κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, ξεκινώ ευχόμενος απλώς καλή χρονιά. Είναι οπωσδήποτε μια χρονιά πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ασφαλώς για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το νομοθετικό αυτό ε, κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι πολύ καλή χρονιά και πολύ καλές εργασίες. Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε με την ιδέα ότι θα μπορούσα να προσφέρω κάτι στις εργασίες της Επιτροπής σας. Το 2017 ήταν ένα έτος πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για το Κοινοβούλιο πάντως, στους τομείς αυτούς, καθώς και υιοθετήσατε την οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας το Μάρτιο, αλλά και εγκαθιδρύσατε, δημιουργήσατε το Σεπτέμβριο την Ειδική Επιτροπή για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ιδιαίτερα λοιπόν με συγκινεί το γεγονό ότι θελήσατε να ακούσετε και τις δικές μας θέσεις. Με την ιδιαιτερότητα που έχουν, ότι δηλαδή η Γαλλία, όπως υπογραμμίστηκε, αφού επλήγει κατά τρόπο αποτρόπαιο και τόσο σοβαρό από την τρομοκρατία, υιοθέτησε ένα ιδιάζων πλέγμα ε, διατάξεων και μέτρων, αρκετά διαφορετικό από αυτό άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ταυτόχρονα, πως με συγκινεί το γεγονό ότι με προσκαλέσατε, γιατί είστε ταυτόχρονα και συμπρόεδρος της ε, Intergroup, της νομοθετικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Παιδιών, μαζί με την κυρία Κινίτσι, είστε συμπρόεδροι. Θέμα των δικών μου, ζήτημα ε, τα και των δικών μου ομοδιοτήτων και που ελπίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα απασχολήσει και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και γενικότερα. Κάθε δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι θα απασχολήσει το θέμα λοιπόν το παιδί όλο και περισσότερο αυτές τις δράσεις πέραν της Διεθνούς Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Παιδιών όπου και τα κράτη-μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση γενικότερα δεν φαίνεται να εκδηλώνουν ιδιαίτερες δραστηριότητες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ε, άρα πιστεύω ότι όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε και προσπιζόμαστε τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ονομάζεται ΕΝΟΚ αλλά και σε επίπεδο ε, Συμβουλίου της Ευρώπης που καλύπτει περισσότερες χώρες και που ιδιαίτερα ε, αποτελεί ένα χώρο συνεργασίας για τα δικαιώματα των παιδιών και ιδιαίτερα των παιδιών τη Γαλλία. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Και χαιρετίζω βεβαίως τους συναδέλφους, τους παλιούς συναδέλφους, πρώην συναδέλφους που βλέπω εδώ και αναγνωρίζω. Και βέβαια το γεγονό ότι είναι εδώ παρόντε μου δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά για την αντιλαγή αυτή των απόψεων. Για την κατάσταση στη χώρα μου, τη Γαλλία, από το 2015 και μετά, αλλά βεβαίως γενικότερα και τη Ευρώπη ολόκληρη, για να μην πω ολόκληρου του κόσμου. Γιατί η κατάσταση είναι ότι εκδηλώνονται πολλές τρομοκρατικέ επιθέσει με πολύ σοβαρέ συνέπειε, εγκαθιδρύεται καθεστώς εκ ανάγκη, εισάγονται διάφοροι αντιτρομοκρατικοί νόμοι, νόμοι για την ενίσχυση της ασφάλειας, μετά ε, από την 1η Νοεμβρίου του 2017 ε, πάβει το καθεστώς εκτάτης ανάγκης και έτσι επανερχόμαστε στο, ε, στην εφαρμογή του κοινού δικαίου για την ασφάλεια για το οποίο θα μιλήσω επίσης και επίσης ήθελα να παρουσιάσω και τις συστάσεις που μπορέσαμε ως προσπιστής των δικαιωμάτων των πολιτών να διατυπώσουμε στο πλαίσιο αυτό. Ο θεσμός πάντως προάσπισης και προαγωγής των θεμελιωδών δικαιωμάτων θα σταθώ στις συνέπειες που μπορεί να φέρουν ε, η νομοθεσία και τα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στα δικαιώματα και της ελευθερίας του ατόμου, που είναι βέβαια και το θέμα, φαντάζομαι, το πρωταρχικό και το αντικείμενο για το οποίο εγκαθιδρύθηκε, συστάθηκε η Επιτροπή σας. Ιδιαίτερος βέβαια στάθηκε και ο Διευθυντής της Υπηρεσίας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα στα ζητήματα αυτά, στην προστασία των δικαιωμάτων, την ανάγκη για τα καταπολέμηση των παραβιάσεων. Υποστήριζω και υπογραμμίζω τα όσα είπε και για τα δικαιώματα των μεταναστών και βέβαια την ανάγκη για εξισορρόπηση, όπως είπε και εκείνος, των μελημάτων για την προστασία της ε, δημόσιας ασφάλειας αλλά και των ελευθεριών. Τι συνέβη λοιπόν στη Γαλλία, τι έχουμε δει από το 2015 στον τομέα της καταπολέμησης τρομοκρατίας. Εν ολίγης. Η τρομοκρατία και κυρίως η εκδήλωσή της τα τελευταία χρόνια μέσω μιας ιδιαίτερου χαρακτήρα και χαρακτηριστικών οργάνωσης φορέα μιας βάρβαρης ιδεολογίας δοκιμάζει τις, τις ε, δημοκρατικές μας χώρες τις αρχές και αξίες τους και ιδιαίτερα το κράτος δικαίου και την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δικαιωμάτων του ανθρώπου που βρίσκονται στο επίκεντρο όλων αυτών των μέσων, των εργαλείων που εκφράζετε και εσείς και εγώ και που αποτελούν τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή χάρτη, συνθήκη για τη λειτουργία, σύμβαση για την διαφύλαξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, αλλά και τις ε, θεμελιώδεις και σταγματικές αρχές που ε, ισχύουν σε κάθε μία χώρα και που συνιστούν το κράτος δικαίου της κάθε μίας χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη Γαλλία συγκεκριμένα από το Σύνταγμα του 1958 με τελευταία του αναθεώρηση του 2008 την ομολογία, τη σταγματική, συγκεκριμένα όσον αφορά τη Γαλλία. Έναντι όλων αυτών και πολύ σωστά το επισήμανε ο Διευθυντής κ. Φλάερτη, το κράτος δικαίου έχει κύριο μέλημα τη διασφάλιση της ασφάλειας, της ασφάλειας, δηλαδή να εξασφαλίσει ότι το θεμελιώδες δικαίωμα στη ζωή, να μην κινδυνεύει κανείς από θανάτωση, από τραυματισμό, από διακινδύνευση της ακαιρεότητάς του της σωματικής, είναι κύριο καθήκον των δημοκρατικών μας κρατών. Και άρα οφείλουν αυτά να αναλάβουν τα μέτρα που απαιτούνται για την προστασία της ασφάλειας των πολιτών με τα εργαλεία και ενδεχομένως ενίσχυση και των εργαλείων για την αντιμετώπιση της τρομοκρατικής απειλής. Πλην όμως, πλην όμως αυτά τα μέτρα, τα θεμητά, μπορούν και να παραβιάσουν τα δικαιώματα ή να θέσουν να τα δικαιώματα και τις ελευθερίες. Γιατί αν κοιτάξουμε τις τελευταίες εξελίξεις, τις ε, μεθόδους ε, παρακολούθηση συλλογής δεδομένων, συλλογής προσωπικών δεδομένων, δημιουργίας ε, αρχείων εθνικών, ε, και βέβαια των αρχείων ε, που προκύπτουν από την οδηγία PNR, την, επιδι... την ε, επιδείνωση του χαρακτηρισμού, την αυστηροποίηση του χαρακτηρισμού των αδικημάτων, την ενίσχυση του ποινικού διατακτικού αλλά και των προληπτικών ιδιαίτερω μέτρων που είναι πολύ περιοριστικά έως και μπορούν να οδηγούν σε αποστέρηση της ελευθερίας και ταυτόχρονα είναι στη διάθεση διοικητικών και όχι δικαστικών αρχών. Όλα αυτά τα μέτρα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης ή ανάπτυξη στη, στα εδάφη των κρατών μας ε, πρόσθετων δυνάμεων τήρησης της τάξης και ασφάλειας ενόπλων ακόμη δυνάμεων στη Γαλλία αλλά και σε άλλες χώρες όπου δεν υπάρχει μόνο η παράδοση της ε, διαφύλαξης της ε, τάξης και ασφάλειας από τις στρατιωτικές δυνάμεις αλλά κυρίως από τις δυνάμεις της αστυνομίας, πολιτικές δυνάμεις αλλά είδαμε ότι έχουμε περάσει αυτό το όριο και έτσι έχουμε τις περιπολίες όπως ονομάζουμε όπως πολιτικές δυνάμεις και βέβαια η ενίσχυση των ελέγχων, ελέγχων και στα σύνορα, ελέγχων και στα μέσα μεταφοράς και βέβαια και η συνεργασία, η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που μπορεί να εκφραστεί με κάποιους περιορισμούς και στην εθνική κυριαρχία. Είναι όλα αυτά τα μέτρα θεμητά, όπως σας τα περιέγραψα. Θεμητά ναι, αλλά θα πρέπει και να διαρωτηθούμε, να ε, γύρουμε ερωτήματα, ερωτήματα που και μένα με έχουν απασχολήσει τα τελευταία δυόμιση χρόνια. αλλά και πολύ νωρίτερα βεβαίως, γιατί ξεκινούμε όχι μόνο με την επιβολή των μέτρων ε, έκτακτης ανάγκης του καθεστώτος ε, περιορισμού των δικαιωμάτων από τον Νοέμβριο του 2015, αλλά και από την ημέρα κατά την οποία τη σήμερα ε, έχουμε σημειώνεται η επέτειος, η τρίτη επέτειος της τρομοκρατικής επίθεσης κατά της σατυρικής εφημερίδας Σαρλί Εμπτώ στις 7 Ιανουαρίου του 2015 και από εκεί ξεκίνησε και βέβαια αναφέρατε και εσείς ε, την νομοθεσία για τη συλλογή πληροφοριών, για τις υπηρεσίες πληροφοριών του 2015, την ε, επεξεργασία της οποίας και εγώ έλαβα μέρος. Ε, όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν με έχουν απασχολήσει και εξεκολουθούν να με απασχολούν. Είναι θεμητά και απαραίτητα δεδομένου του νομοθετικού πλαισίου που υφίσταται. Τα μέτρα αυτά δηλαδή τα οποία λαμβάνονται και εισάγονται προσθέτουν κάτι περισσότερο ή έχουν μόνο πολιτικό χαρακτήρα. Είναι πράγματι αποτελεσματικά τα μέτρα αυτά. Και πάνω απ' όλα, και αυτή άλλωστε είναι και η φιλοσοφία που σας εξέθεσε ο κύριος Φλάιρτη και πολύ σωστά, ε, οι επιθέσεις κατά αυτών των αξιών μας, των ελευθεριών μας, από τον τρομοκράτη που θέλει να καταρρύψει τις δημοκρατίες μας, μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα περιοριστικά της ελευθερίας. Δηλαδή πρέπει να περάσουμε στο πεδίο πάνω στο οποίο ακριβώς εντοπίζεται η επίθεση και να το αμφισβητήσουμε ή πρέπει να διαφυλάξουμε ζηλότυπα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας εκδηλώνοντας την παρησία, γιατί περί αυτού πρόκειται την παρησία να αγωνιστούμε με τα δικά μας τα όπλα, που είναι τα όπλα της ελευθερίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Δεν θα παραθέσω τα δικά μου λόγια, αλλά τα λόγια του Προέδρου του Σταγματικού Συμβουλίου της Γαλλίας, του Λορόν Φαμπιούς, ο οποίος το 2016 έλεγε ότι ενισχύοντας τα μέτρα ασφάλειας ε, για λόγους υποτιθέμενης ασφάλειας ε, κινδυνεύουμε να ενισχύσουμε τους ίδιους τρομοκράτες. Έτσι λοιπόν, ο αγώνα κατά τη τρομοκρατία θα πρέπει να διεξάγεται και σε εθνικό αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσα από το σεβασμό των δικαιωμάτων των αρχών τη Ευρώπη, δηλαδή δικαιώματα, προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών και αυτή είναι η ευθύνη του καθενό από εμά και συγκεκριμένα στο άρθρο 23 τη Οδηγία για την καταπολέμηση τρομοκρατία προ το τέλο ε, του κειμένου τη Οδηγία, του διατακτικού, αναφέρεται ξεκάθαρα στο άρθρο 23 ότι τα μέτρα τα οποία έχει περιγράψει η Οδηγία πρέπει να λαμβάνονται μέσα στο, σε, σε σεβασμό, σε συνθήκε σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και ε, της οδηγίας της 15 Μαρτίου του 2017. Ε, το ξέρουμε πολύ καλά και η Γαλλία το έζησε ότι η κοινή γνώμη, η συγκνησιακή φόρτιση και είμαι και εγώ όπως ο καθένας σας φοβάμαι, φοβούμαστε όλοι και μετά τρομοκρατικές επιθέσεις και πριν από μια τρομοκρατική επίθεση και ο καθένας πάντα διαρωτάται πότε μπορεί να ξαναεκδηλωθεί μια τέτοια επίθεση. Και οι αρχές μας λένε ότι η απειλή είναι παρούσα, σε πολύ ψηλό επίπεδο, παρούσα. Είναι πίεση λοιπόν αυτή της κοινή γνώμης αλλά και της κινησιακής φόρτισης και έτσι τα κράτη-μέλη είναι έτοιμα να εισαγάγουν νέα μέτρα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας που περιορίζουν ακόμη περισσότερο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες χωρίς να ε, κάνουν διάκριση στις χώρες μας, ιδιαίτερο στη Γαλλία, αλλά σε όλες τις χώρες. Ας κοιτάξουμε τι συμβαίνει στη Δανία, το Βέλγιο, τις κατοχώρες, την Ισπανία, την Ιταλία, τη Γερμανία. Σε όλες μας τις χώρες, λοιπόν, δεν γίνεται πραγματική συζήτηση για το θέμα. Γιατί η κοινωνία αισθάνεται τέτοιο φόβο και τέτοια αγκύλωση που τα μέτρα που έχουν χαρακτήρα ενίσχυσης ασφάλειας, ενίσχυσης ασφάλειας αλλά όχι προστασίας τόσο των ελευθεριών, την χάνουν ομόφωνης ή σχεδόν ομόφωνης υποστήριξης και μάλιστα ορισμένοι πλειοδοτούν κιόλα υπέρ ακόμη περισσότερη ασφάλεια. Και το είδαμε και στη συζήτηση στα κοινοβούλια, στο άρθρο 8, παραδείγματι, ενό νόμου της 30 Νοεμβρίου, 3, 3 Ιουλίου του 2016 συγκεκριμένα, με ένα κείμενο λοιπόν το οποίο αναφερόταν στη δυνατότητα να ε, κρατηθεί κάποιος για ορισμένε ώρες, να προσαχθεί και να κρατηθεί χωρίς παρέμβαση εισαγγελική κτλ. Και έγινε συζήτηση για 4-5 ώρες. Και αυτή ήταν η μόνη συζήτηση που έγινε μέσα στο Κοινοβούλιο μεταξύ διαφόρων βουλευτών που αντιπαρέθεταν τις απόψεις τους. Στην προηγούμενη ε, Βουλή της Γαλλίας το προηγούμενη, ε, στα προηγούμενα δεδομένα πλειοψηφίας, δηλαδή με πλειοψηφία σοσιαλιστική και αντιπολίτευση από τη δεξιά. Και το μόνο επιχείρημα έναντι αυτών οι οποίοι ήταν κατά των μέτρων που προβλήθηκε ήταν ότι αγαπητοί συνάδελφοι, αν κάνουμε αυτό που λέτε και δεν υιοθετηθεί αυτό το μέτρο, δέχεστε εσείς να αναλάβετε την ευθύνη αύριο κάποιος τρομοκράτης, άντρας ή γυναίκα, να μπορέσει, ακριβώς επειδή δεν ετέθησε σε εφαρμογή το μέτρο της ε, κράτησης για τέσσερις ώρες, γιατί αυτό ήταν το μέτρο, να ε, προχωρήσει σε τρομοκρατική πράξη. Τι ευθύνη αναλαμβάνεται εναντί των πολιτών, εναντί των Γάλλων. Καταρρυπτικό το επιχείρημα. Προφανώ ένα σύστημα δημοκρατικό που κανεί κοιτάει να ξαναεκλέγει, γιατί σε ένα δικτατορικό σύστημα δεν χρειάζεται να το συζητήσει, αλλά σε ένα δημοκρατικό σύστημα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου συζήτηση και διάλογο όπω αυτό που γίνεται εδώ στην Επιτροπή σα, οι θέσει που εγώ ε, υιοθέτησα, είναι πολύ δύσκολο όχι να εκφραστούν τόσο όσο να γίνουν κατανοητές. Γιατί επικρατεί η ιδέα ότι πρέπει να πράξουμε το άπαν και όταν λέω το άπαν εννοείται ότι δεν με νοιάζει καθόλου για την προστασία, για τις εγγυήσει ε, ανθρωπινών δικαιωμάτων κτλ. Πρέπει να πράξουμε το άπαν για να προληφθεί και βεβαίως να κατασταλεί αν τυχόν ε, ο ΙΜΕ διαπραχθεί μια τρομοκρατική ενέργεια. Έτσι έγιναν τα πράγματα στη Γαλλία. Έτσι συνέβη και έτσι όντως μέσα από αυτό το πνεύμα προχωρήσαμε μετά τις 13 Νοεμβρίου, συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου το 2015, γιατί ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αποφάσισε, είχε και την σχετική εξουσία δυνάμει του νόμου, με διάταγμα προεδρικό, το οποίο ε, υπέγραψε τη νύχτα της 13ης προς 14η μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις που έλαβαν χώρα γύρω στις 10-11 το βράδυ 13 ε, Νοεμβρίου στο Παρίσι έλαβε την απόφαση και εγκαθίδρυση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και έτσι φτάσαμε να πραγματοποιήσει η Γαλλία ε, ένα 11 το βραδυ 13 άνευ προηγουμένου, συγκεκριμένα μόνο η Γαλλία, όχι άλλα κράτη, με την εγκαθίδρυση αυτού του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης, ε, το οποίο και καθεστώ έλαβε παράταση πέντε φορές, με νόμους αυτή τη φορά, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου του 2017. Επικράτησε δηλαδή το καθεστώς αυτό επί περίπου δύο χρόνια, ενώ το καθεστώς εκτά της ανάγκης είναι εξορισμού εξαιρετικό και προσωρινό μέτρο. Κατά την περίοδο αυτή, το υπενθυμίζω και είναι πολύ σημαντικό, έγινε επίκληση και χρήση του άρθρου 15 τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, δηλαδή εμεί είπαμε ω Γαλλία στο Συμβούλιο τη Ευρώπη ότι ήμασταν σε θέση να λάβουμε μέτρα τα οποία απέκλειναν από ορισμένα άρθρα τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Όμω από 1η Νοεμβρίου του 2017 πλέον αυτό δεν ισχύει, δηλαδή πλέον επαναρχόμαστε στη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Άρα ό,τι έχω να σα πω από εδώ και πέρα, από την 31η Οκτωβρίου και μετά, οφείλει να σέβεται την ε, Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης και επιπλέον η Γαλλία με την απόφαση αυτή της 3ης Ιουνίου, λέει τώρα πρόεδρος του 2015, υιοθέτησε αυτά μέτρα και χαρακτηριστικό είναι ότι στα κείμενα αυτά και η σχετική νομοθεσία που υιοθετήθηκε μέσα σε ένα συγκεκριμένο κλίμα, όπως σας είπα, και ως εκ τούτου τα μέτρα αυτά δεν εξετάστηκαν ως προς την συνταγματικότητά τους πριν να υπογραφούν και να δημοσιευθούν από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 60 βουλευτές και 60 γερουσιαστές δηλαδή ε, από το, η Βουλή και τη Γερουσία, από τη και τη Γερουσία, δεν προσέφηγαν στο Συνταγματικό Δικαστήριο για να ζητήσουν την εξέταση της συνταγματικότητας των μέτρων αυτών. Κλείνω την παρένθεση και αυτό έχει σαν συνέπεια ότι η συνταγματικότητα των μέτρων αυτών εξετάζεται μόνο κατά περίσταση, μήνα το μήνα, μέσω μιας διαδικασίας η οποία μάλιστα ε, προβλέπεται από την αναθεώρηση του 2008, δηλαδή μια ε, ρήτρα εξέταση ταχματικότητας που έχουν και άλλες χώρες βεβαίως και άλλες τάξεις, που σημαίνει παρεμπίπτουσα εξέταση κατά τη διάρκεια μιας άλλης δίκης ενώπιον ενό οποιοδήποτε άλλου δικαστηρίου με επίκληση συνταγματικότητα ή ένσταση συνταγματικότητα καλύτερα. Οπότε διακόπτεται η δίκη και πάμε στο συνταγματικό δικαστήριο, το οποίο πρέπει να εξετάσει εάν η διάταξη στο σταγματικο οποία ε, πρόκειται να εφαρμοστεί ή να εξεταστεί η εφαρμογή της από το ε, κύρια δίκη είναι σταγματική ή όχι. Και έτσι έχει γίνει επίκληση σταγματικότητας από ε, διάφορες, ε, σε διάφορες περιστάσεις, δυνάμει μάλιστα και της νομοθεσίας του 2013 της, για την καταπολέμηση της δημοκρατίας και αποδεικνύεται ή κρίνεται κατά περίσταση και παρεμπιπτόντως ότι ήταν αντισταγματικά τα μέτρα αυτά. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά Εδώ έχουμε και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι δεν προβλέπεται στο Σύνταγμά μας και μάλιστα προσπάθησε η κυβέρνηση να ενσωματώσει στο Σύνταγμα, αλλά δεν προβλεπόταν η διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος, δεν ολοκλήρωσε, δεν έφτασε στο σκοπό της καλύτερα, διότι συνδέθηκε με την εγγραφή σε συνταγματικούς όρους με την αναθεώρηση του καθεστώς έκτη ανάγκης και ταυτόχρονα την δυνατότητα για αποστέρηση της ηθαγένειας από πολίτες που είχαν διπλή ηθαγένεια. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μία κύρια αρχή, σε σχέση με την ηθαγένεια για τη Γαλλική Δημοκρατία. Τα δύο αυτά δηλαδή ζητήματα οδήγησαν σε αυτά τα αποτελέσματα, ότι δηλαδή δεν ενεγράφει στο Σύνταγμα με νόμο, απλό νόμο του 1955 προβλεπόταν αυτό. Ένας νόμος ο οποίος είχε υιοθετηθεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του, ε, του Αλγερικού όπως ονομαζόταν τότε, τώρα ονομάζεται πόλεμος της Αλγερίας. Πρόκειται για ένα καθεστώς το οποίο εν ολίγης σημαίνει ότι οι διοικητικέ αρχές, η διοικητική αρχή έχει τη δυνατότητα να αναλάβει κάποια μέτρα περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα τα οποία εκτός καθεστώτος της ανάγκης είναι μέτρα που μπορεί μόνο ο δικαστής να επιβάλλει. Ενώ στην περίπτωση αυτή νομάρχης, διοικητική αρχή, ε, αστυνομική αρχή μπορεί να επιβάλλει περιοριστικά της ελευθερίας μέτρα, ε, κατοίκο περιορισμό, ε, κλείσιμο χώρων λατρείας, ελέγχους ταυτότητας, ελέγχους αποσκευών και ούτω καθεξής. Αυτό είναι εν ολίγης το σύστημα των έκτακτων μέτρων που έχει στη διαθεσή της η διοίκηση, οι διοικητικές αρχές δυνάμει αυτής της διατάξεως. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μέτρα τα οποία έχουν προσωρινό χαρακτήρα και προσωρινό λοιπόν χαρακτήρα και περιορισμένο χαρακτήρα γιατί παρεμ παραβιάζουν ή περιορίζουν το άρθρο 60 του συντάγματός μας που όμως έχει αντίστοιχα και σε άλλα ε, συνταγματικές ε, τάξεις για τις ατομικές ελευθερίες που ορίζει δηλαδή ότι οι ατομικές ελευθερίες την χάνουν προστασία από τον δικαστή, από τη δικαστική αρχή και ότι μόνο δικαστική αρχή έχει εξουσία για αποστέρηση κάποιων πολιτών από τις ελευθερίες τους και όχι η διοίκηση ή κάποια διοικητική αρχή. Βεβαίω και παράλληλα με αυτό καθιστώ σε κράτη ανάγκη. θα το εκθέσω και αργότερα, ακολούθησε μια σειρά διατάξεων του λεγόμενου κοινού δικαίου που παραμενουν ισχυ ενισχύει. Δηλαδή, από 1η ε, Νοεμβρίου του 2017 πάβουν να ισχύουν κάποια έκτακτα μέτρα και διατάξεις, άλλα όμως που είτε προϋπήρχαν είτε θεσπίστηκαν με την, με το καθώς της ανάγκης παραμένουν ενισχύ. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προβληματιστούμε εάν τώρα που πλέον δεν ε, ισχύει το άρθρο, δεν υπάρχει επίκληση του άρθρου 15 της Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, μπορούν ακόμη να είναι συμβατά με την Σύμβαση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων του ε, Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης, κυρία Πρόεδρε, και δεν θέλω να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες βεβαίως, αλλά ρωτήσατε τι κάναμε τι κάναμε λοιπόν. Εκφράσαμε και εκφράσαμε με επιμονή και επανειλημμένο τις επιφυλάξεις και τους προβληματισμούς μας, αντίθετα στο ρεύμα βεβαίως, αντίθετα στο ρεύμα της κοινή γνώμης, αντίθετα στο ρεύμα της πολιτικής τάξης που εξέφρασε την πλειοψηφία. Επίμονα και επανειλημμένα υπογραμμίσαμε ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ του θεμητού μελήματος για ασφάλεια και του σεβασμού και των εγγυήσεων για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Και υπογραμμίζαμε ότι δεν είναι δυνατόν η πλάστη να υπερβολικά προς την πλευρά της ασφάλειας. Και έτσι, με την υιοθέτηση για την αντικατάσταση καθώς της ανάγκης ενός νόμου που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως νόμος υπερβολικής ε, δημόσιας τάξης και ασφάλειας στις 30 Οκτωβρίου 2017 επιλέγει η γαλλική κυβέρνηση να δώσει περισσότερη έμφαση στην ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, στην ενίσχυση της ασφάλειας, δηλαδή ανατρέπει αυτή την ισορροπία. Ταυτόχρονα, έχοντας δει και ε, τις προσφυγές και παρατηρήσεις των θυγωμένων από αυτά τα μέτρα, περί τις 600. Τις μελετήσαμε και είδαμε πολλές περιπτώσεις ε, πολιτών και γενικότερα περιορισμού κατοίκων και αποστέρησης ελευθεριών. Πρόκειται για ζητήματα που αφορούσαν, με δεοντολογικά ζητήματα στη συμπεριφορά των αστυνομικών δυνάμεων, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι έρευνες κατοίκων από τις αστυνομικές αρχές. Δώσαμε απάντηση στα, στις προσφυγές αυτές με δύο τρόπους. Πρώτον, διατυπώνοντας ε, συστάσεις για την εφαρμογή των μέτρων αυτών σε σχέση με τις κατοίκων έρευνες παρουσία ανηλίκων όπου επισημάνομαι ότι χρειάζεται να λαμβάνονται κάποια προληπτικά μέτρα και βέβαια και το Συμβούλιο της Επικρατείας και οι διοικητικές αρχές ακολούθησαν αυτές τις συστάσεις και προτάσεις. Υιοθετήσαμε συστάσεις σε σχέση με την διεξαγωγή των ερευνών κατοίκων σε σχέση με τα πρακτικά ε, της κατοίκων έρευνας που πρέπει να παραδίδεται, να παραδίδονται στον ενδιαφερόμενο, στην αποζημίωση που πρέπει να προκύψει ε, για όποια ζημία έχει προξενήσει μια ε, κατοικονέρευνα και με μια απόφαση της 6ης Ιουλίου το Συμβούλιο της Επικρατείας ακολουθεί μια πιο θετική και ευνοϊκή θα έλεγα ως προς την αποζημίωση ε, ζημίας του πολίτη που ξεπερνά την προϋπόθεση της ε, βαριά αμέλεια όπω ίσχυε προηγουμένω, που ήταν πολύ δύσκολο να αποδειχθεί. Επίση, ε, ο κατοίκον περιορισμό. Με μια κατάφορη περίπτωση ενός καθηγητή του Λυκείου που είχε ε, στον οποίο είχε, αποκλεισ... είχε επιβληθεί κατοίκον περιορισμός για τις ώρες που θα έπρεπε να είναι στο μάθημά του. Μπορέσαμε να το αμφισβητήσουμε αυτό για να του επιτρέπεται η μετάβαση στο σχολείο για τις ώρες των μαθημάτων. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια περίοδο βέβαια χρονική όπου ελήφθη μεγάλος όγκος τέτοιου είδους αποφάσεων γύρω από τα γεγονότα του Νοεμβρίου του 2015. Επίσης πέρυσι, Μάιο-Ιούνιο, υιοθετήσαμε μια απόφαση που ίσως ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και θελήσει να τη μελετήσει. Μια απόφαση που έχει να κάνει με την ε, παροχή φροντίδας και αποζημίωση των θυμάτων της τρομοκρατίας και ξέρω ότι εδώ υπάρχουν βουλευτές που ιδιαίτερα μεριμνούν για τα ζητήματα αυτά και έτσι εδώ ιδιαίτερα μας απασχόλησε και προτείναμε μια σειρά μέτρων αποζημίωση των θυμάτων. Ε, μιλήσαμε επίσης για τα εις ζημίες των μέτρων αυτών. Φερρυπίν, κάποιος που ε, γίνεται αντικείμενο έρευνας κατοίκων και άνθρωπος του περιγύρου του, του οικογενειακού του κύκλου, ε, μπορεί να απολυθεί γιατί ε, έχει γεννήσει υποψίες στον διευθυντή του. Αυτό λοιπόν το αντιμετωπίζουμε. Και επίσης, για να τελειώσω, χρησιμοποιήθηκαν τα μέτρα αυτά έκτακτης ανάγκης, για να μην πω καταστρατηγήθηκαν, για να πραγματοποιηθούν επιχειρήσεις διατήρησης της τάξης, δηλαδή συλλογικά και ατομικά μέτρα του καθεστώτος και της ανάγκης, αξιοποιήθηκαν χωρίς να έχουν άμεση συνάφεια με την τρομοκρατική επιλή για να εξασφαλιστεί παρέμβαση σε περίπτωση διαδηλώσεων. Ξέρεις να θυμάστε συγκεκριμένα τον, ε, την άνοιξη του 2016 με το ε, εξάμεινο για να πω πέντε μήνες ε, εκείνο των διαδηλώσεων που είχαν να κάνουν με την αναθεώρηση του εργατικού κώδικα, τη λεγόμενη νομοθεσία, το λεγόμενο νόμο Ελκομρή από το όνομα της Υπουργού Εργασία την εποχή εκείνη. Και για να ολοκληρώσω μετά το καθεστώ εκτάκτη ανάγκη, πώς έχουν τα πράγματα τώρα. Εδώ τώρα πια έχουμε να κάνουμε με το νόμο της 30 Οκτωβρίου 2017, νόμο με τον οποίο τίθεται τέρμα στο καθεστώ εκτακτής ανάγκης, αλλά ταυτόχρονα εισάγεται μια σειρά μέτρων για τα οποία η κυβέρνηση δηλώνει η ίδια η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα έχουν αποτέλεσμα ισοδύναμο με αυτά του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης. Και έτσι, αυτός ο νόμος της 30 Οκτωβρίου εισάγει στο κοινό δίκαιο πλέον το, ε, μια σειρά διατάξεων που προκύπτουν από το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, το, η περάτωση του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης πλέον είναι μόνο μία θεωρητική ε, κατασκευή. Έχουμε να κάνουμε με ε, έλεγχο στην πρόσβαση και την κυκλοφορία των ε, προσώπων, επαλήθευση ταυτότητας, έλεγχο σωματικό, έλεγχο αποσκευών σε διάφορες, σε διάφορες περιμέτρους ασφαλείας όπως αυτές μπορεί να χαρακτηριστούν γύρω από χώρους εκδηλώσεων, κλείσιμο χωρών λατρείας που πέρασε πλέον από το καθώς ανάγκης στο κοινό δίκαιο και σε μια διατύπωση που μας απασχόλησε και μας ανησύχησε ιδιαίτερα ότι δηλαδή εάν ιδέες ή θεωρίες ε, που εκφράζονται μέσω των λόγων ή δραστηριότητε ε, που μπορούν να οδηγήσουν σε ανησυχίες για την τρομοκρατία κτλ. τότε επιλαμβάνεται η σχετική αρχή. Εμένα προσωπικά με απασχόλησε ιδιαίτερα το γεγονός αυτό και το να εξετάσω εάν μια ε, ιδέα ή θεωρία μπορούσε να οδηγήσει σε αυτό που παλαιότερα, σε παλαιότερη νομοθεσία χαρακτηριζόταν ως έγκλημα σχετικό με την έκφραση άποψη γνωμης Άρα δηλαδή, όταν και εντό εισαγωγικών το λέω, υπάρχουν ανησυχίες σοβαρές ότι η συμπεριφορά ενός ατόμου μπορεί να αποτελεί σημαντική απειλή για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη, κλείνουν τα εισαγωγικά. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ ασαφή διατύπωση και ευρύτατη δυνατότητα ερμηνείας του τι σημαίνει σοβαρές ανησυχίες ή κίνδυνοι που οδηγούν εν τέλει στην δυνατότητα εισαγωγής αυστηρότατων ε, και σοβαρότατων ελέγχων και περιορισμών των ελευθεριών, ε, κατοίκων περιορισμός, υποχρέωση για παρουσία και ε, έλεγχο από τις αρχές, απαγόρευση κυκλοφορίας, απαγόρευση επικοινωνίας με συγκεκριμένα άτομα και επίσης εν τέλει αυτό που ονομάζεται στην νομοθεσία επίσκεψη και δημεύση, αυτό που παλαιότερο ονομαζόταν ε, διοικητική έρευνα, από διοικητικές αρχές δηλαδή, που είχε χαρακτήρα ε, προστατευτικού μέτρου, δηλαδή ότι προληπτικά πριν από την ε, επίσκεψη για την, κατοίκο, για την έρευνα απαιτούνταν η άδεια από δικαστική αρχή, αλλά τώρα πλέον οι προθεσμίες που έχουν επιβληθεί καθιστούν αδύνατη αυτή την έγκριση. Γιατί στην πραγματικότητα θα πάει η αρχή στον δικαστή, θα του δώσει ένα χαρτί και όπως λεγόταν και στις συζητήσεις, όπως είπα νωρίτερα στο Κοινοβούλιο, θα του πει αν δεν μου δώσετε την άδεια κύριε δικαστά αμέσως για αυτή την κατοίκον έρευνα, θα είναι αργά πια και τι είδου ευθύνη μπορείτε εσείς να αναλάβετε. Αυτή είναι η κατάσταση και έτσι έχει διατυπωθεί ο νόμος. Επιπλέον, και όπως είπαμε, έχουμε τώρα ένα πλέγμα νομοθετικό το οποίο σε μεγάλο βαθμό αντιγράφει αυτά τα οποία προέβλεπε και το καθεστώς της τη Και επιπλέον, και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ε, ε, γύρεται το ζήτημα της συνταγματικότητας ή της συμβατότητας με το Σύνταγμα αυτών των διατάξεων και θα συνεχίσει να τίθεται, γιατί ο προσωρινό ή χαρακτήρας χαρακτήρα ε, των μέτρων ε, σημαίνει διαφορετική αξιολόγηση σε σχέση με τα θεμελιώδη δικαιώματα και υπάρχει και μια άλλη σειρά νομοθετημάτων που σας εξέφασα και νωρίτερα που ενισχύουν το πλέγμα των νομοθετικών διατάξεων, μια σειρά από διατάξεις για την πρόληψη της τρομοκρατίας, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, ενισχυμένη, διοικητικός έλεγχος, έλεγχος από τις διοικητικές αρχές των προσώπων που ε, ε, επανέρχονται από επίσκεψη στο εξωτερικό, όταν και αναφέρεται έτσι. Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ε, που οδηγούν σε μελήματα για το κατά πόσον μπορεί να έχει έρθει σε επαφή με τροποκρατικές ομάδες και ως συνέπεια να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια του συγκεκριμένου πρόσωπου. Καταλαβαίνετε τι ευρύ περιθώριο ερμηνείας και δράσος υπάρχει εδώ και βεβαίως η περίφημη αυτή κράτηση για τέσσερις ώρες που σας ανέφερα νωρίτερα, του νόμου της 3ης Ιουνίου. Πάλι με αιτιολόγηση ότι υπάρχουν σαφείς ε, ε, λόγοι να υποπτεύεται κανείς ότι μπορεί να έχει συνάφεια με τρομοκρατικές ε, δράσεις στο συγκεκριμένο άτομο όλο, εμείς θεωρούμε ότι ε, η επιχειρηματολογία που λέει ότι δεν παραβιάζουν τις ελευθερίες τα κείμενα αυτά και οι διατάξεις αυτές γιατί έρχονται να δώσουν απάντηση σε μια άκρος έκτακτη κατάσταση, μια άνευ κατάσταση, δηλαδή την τρομοκρατία, για μας δεν ευσταθεί, διότι σε καμία περίπτωση δεν περιγράφεται τι ακριβώς είναι η τρομοκρατία, δεν υπάρχει ορισμός της τρομοκρατίας και βεβαίως εδώ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου, και νομίζω ότι αυτό είναι το δίδαγμα που πρέπει να αποκομίσουμε, βρισκόμαστε σε μια κατάσταση λοιπόν όπου από το τέλη του 2015 έχουμε μπει σε μια λογική υποψίας. Δηλαδή, στο ποινικό δίκαιο και τα δικηματά του έχουμε αξιολόγηση όχι από πράξεις ή συμπεριφορά συγκεκριμένη, από συγκεκριμένο δείγμα που έχει διαπραχθεί, αλλά απλώς και μόνο και όπως είπα στηριζόμενοι μόνο σε υποψία, αξιολόγηση προσωπικότητας, αξιολόγηση συμπεριφοράς σε μια συγκεκριμένη κατάσταση. Και όπως είπα και εγώ νωρίτερα από τον Ιανουάριο του 2016 σε μια ε, συνέντευξή μου στην εφημερίδα Le Monde, είχα επισημάνει και μια και είχα κάνει και ένα παραλληλισμό με την περίοδο της, του τρόμου ε, μετά τη Γαλλική επανάσταση ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε μια τέτοια κατάσταση και το επανέλαβα και τον Ιανουάριο του 2017 ότι βεβαίως πρέπει να έχουμε ενισχυμένη δράση για την καταπολέμηση τρομοκρατίας αλλά ε, το να αποκοπεί αυτό από την τιμώρηση για να μετατραπεί η καταπολέμηση τρομοκρατίας σε ένα μέτρο καταστολής μετατρέπει την κοινωνία μας από κοινωνία ευθύνη σε κοινωνία κάχη υποψίας και υποψίας και έτσι κάθε υπετιότητα ε, βγαίνει από το εξεταζόμενο πλαίσιο, επιβάλλονται μέτρα κατασταλτικά με το διοικητικό και το ποινικό δίκαιο και έτσι αποκόπτεται κάθε ε, συνάφεια από την ε, έννοια της διάπραξης ενός εγκλήματος και μετατρέπεται σε αξιολόγηση επικινδυνότητας. Δηλαδή ε, χάνεται πλέον η διάκριση μεταξύ ανθρώπου και μη ανθρώπου και βέβαια χάνεται και το τεκμήριο της αθότητας. Και ένα παράδειγμα σε αυτά είναι η αναγνώριση ενός ε, αδικήματος σε ε, σελίδες που έχουν να κάνουν με την ε, έκφραση υποστήριξη στην τρομοκρατία, που δύο φορές ακυρώθηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί είπε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί το Σύνταγμα προκειμένου ένα τέτοιο αδίκημα να υλοποιηθεί πραγματικά. Ε, πρέπει να αντλήσουμε το εξής δείγμα ότι πρέπει να αποκοπούμε τις, ε, από τις ε, νομικές εξηγήσεις του ζητήματος όταν μιλούμε για την νομιμότητα δηλαδή των αξιόπινων πράξεων δηλαδή χρειάζεται να είναι προβλέψιμος ο ορισμός και επίσης να έχουμε και την σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των δικαστικών διατάξεων για αυτές τις αξιόπινες πράξεις. Ε, πλέον έχουμε εκφύγει αυτής της νομικής ε, σαφήνειας ε, και έτσι αποδυναμώνουμε το κράτος δικαίου. Και θα ολοκληρώσω, Πρόεδρε, λέγοντας πως στις χώρες μας τη σήμερα ημέρα ε, αντιμετωπίζουμε ένα διτό οικοδόμημα ε, ποινικού δικαίου, του τακτικού ποινικού δικαίου και του τρομοκρατικού ε, ποινικού δικαίου που ε, έχει μετατραπεί σε ένα ε, ποινικό διοικητικό δίκαιο που επιτρέπει να λαμβάνονται μέτρα που δυνάμει μπορούν να περιορίσουν τις προσωπικές ελευθερίες και τα δικαιώματα. Οι διατάξεις του νόμου ε, του, της 30 Οκτωβρίου 2017 δεν ε, περιέχονται στον ποινικό κώδικα, αλλά στον κώδικα της εσωτερικής ασφάλειας. Ε, δηλαδή, απομακρυνόμαστε από τα κείμενα που εφαρμόζει το δικαστικό σώμα και πλησιάζουμε την νομοθεσία τη επιβολή του νόμου που εφαρμόζει η υπηρεσία πληροφοριών, που εφαρμόζει η αστυνομία. Και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, διότι αυτή η ε, κατάσταση δεν σημαίνει μόνο σε εμά. Ε, μην ξεχνάμε το Terrorism Act του 2000 ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προβλέπεται για τις αρχές επιβολής νόμου ευρύτατη αρμοδιότητα παρεμβαίνουν με ανακρίσεις, με κατασχέσεις, με οτιδήποτε θέλουν στα σύνορα, στα λιμάνια για την δίωξη τρομοκρατικών ενεργειών χωρίς πρώτερη έγκριση, χωρίς να υπάρχει βάσιμη υποψία για τρομοκρατική ενέργεια. Επίση, με τα βιομετρικά δεδομένα μπορούν να κατεβάσουν τα περιεχόμενα ολόκληρου του τηλεφώνου ε, και ε, γι' αυτό και ε, υπάρχει η υπόθεση κατά του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, αυτά, Πρόεδρε. Ε, όλα αυτά εγγράφονται στα πλαίσια ενισχυμένης συνεργασίας ε, κάποιων κρατών μελών και ενδεχομένως ε, στη συνέχεια να τοποθετηθώ και για αυτό το, που, το θέμα που θίξατε για την διαλειτουργικότητα, έτσι την πρόταση της 12 η Δεκεμβρίου της Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Συνεργαστήκαμε με κράτη-μέλη στη διάσκεψη που έγινε το Σεπτέμβρη του 17 ε, στο Στρασβούργο, στα πλαίσια του ΛΥΠΚΑΝ, είναι ένα άτυπο πλαίσιο, 15 ε, περίπου οργανισμοί που ασχολούνται με τα διοντολογικά ζητήματα των συστημάτων ασφαλείας, η Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, διάφορες μεγάλες χώρες εκπροσωπούνται και το Βέλγιο. Ε, σε αυτή τη διάσκεψη λοιπόν ε, συγκρίναμε τις εμπειρίες μας και προσπαθήσαμε να μελετήσουμε αυτό το ζήτημα. Ξυπακούεται ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί η ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια ε, και την ελευθερία και απευθύναμε επίκληση προς τις ε, ευρωπαϊκές αρχές, ε, γενικότερα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να θεσπιστούν εξωτερικοί μηχανισμοί ελέγχου των αρχών ασφαλείας, ούτως ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι εταίροι να μπορέσουν να διαβουλευτούν και καταλήξουν σε κάποιες, συγκεκριμένε σε κάποιες συγκεκριμένες διατάξεις, λοιπόν. Πρόεδρε, Σήμερα το απόγευμα θα σας έλεγα ότι είναι θεμητός ο στόχος. Ναι, πρέπει να σώσουμε τις ζωές πολλών αντρών, γυναικών, παιδιών. Ναι, πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτές τις βάρβαρες ε, τρομοκρατικές οργανώσεις, ε, οργανώσεις ανίποτης ε, βαρβαρότητας. Πρέπει να τις καταπολεμήσουμε γιατί κινούμεθα σε ένα δικαστικό αστυνομικό πλαίσιο που δεν γνωρίζει ουσιαστικά σύνορα και γι' αυτό από κοινού θα πρέπει να κινηθούμε σεβόμενοι τις αρχές του κράτους, του δικαίου, βασικές ελευθερίες και τα βασικά δικαιώματα, πιστεύω πώς αυτή είναι η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να την επομιστεί, να την επομιστείτε όταν θεσμοθετείτε, όταν νομοθετείτε, συγγνώμη. Ε, σήμερα, αύριο, ε, για τα νομοθετήματα που εξεργάζεστε μέχρι, ε, σε όλη την περίοδο μέχρι το Σεπτέμβριο. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ασκήσει την επιρροή της επί των κρατών μελών. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να σεβαστούν αυτά τα δικαιώματα, διότι πρόκειται για εθνική κυριαρχία ε, και η εθνική κυριαρχία, όποιες και ας είναι οι ενωσιακές ε, πολιτικές ε, από τον καιρό του τρίτου πυλώνα, όπως έλεγε ο κύριος Σοφλάιρτη, ό,τι και να έχει συμβεί, πρόκειται για θέματα εθνικής κυριαρχίας. Χρειαζόμαστε μηχανισμό ελέγχου, ο οποίος μηχανισμός ελέγχου όμως προς το παρόν ε, κινείται σε εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό ζητώ εξωτερικό έλεγχο. Είναι απαραίτητο, είναι το νον ουκάνευ αυτό ο μηχανισμό. Δεν γίνεται να διατηρήσουμε αυτή την νομιμοποίηση εάν δεν ε, πληρούμε αυτή ε, την εγγενή υποχρέωση σεβασμού του κράτου δικαίου των βασικών ελευθεριών και επιμονή μου βάσεως ε, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος των αρχών. Επιμονή μου βάσεως να, να προσέχουμε να μην ε, διέρχονται αυτή την ε, κίτρινη γραμμή, ούτε καν την κόκκινη, την κίτρινη γραμμή τα κράτη-μέλη. Και ελπίζω σε αυτό το διάλογο να συνέβαλα με αυτή την παρέμβασή μου. Ε, κύριε Τομπόν, ναι, μπορούμε να σας χειροκροτήσουμε νομίζω, διότι ε, με εκπληκτικό ε, αριστοτεχνικό τρόπο θέσατε το δάκτυλο επί του τύπου των ύλων ε, και μας παρουσιάσατε νέες απειλές που ε, υποθάλπονται από ε, ανθρώπους ε, που γνωρίζουν δυστυχώς εκ των έσω τα συστήματα ασφαλείας μας. Εξαιρετική η παρουσίαση που κάνατε του γαλλικού συστήματος που από όλα τα ευρωπαϊκά συστήματα είναι αυτό που γνωρίζει τη μεγαλύτερη απειλή, είναι καθημερινή απειλή, εξαιρετικά υψηλή. Και Γι' αυτό το λόγο έχει θεσπίσει μια σειρά ε, εργαλείων. Μιλήσατε για το, ε, το καθεστώς έκτακτης ανάγκης. Το τι συνεπάγεται αυτό και όταν μιλήσατε για την νομιμοποίηση, ναι, είπατε ότι νομιμοποιείται ο στόχος, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να γίνει σεβαστό το κράτος δικαίου και να διατηρείται η ισορροπία. Επίσης, ε, απευθύνεται επίκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Επιτροπή μας ε, μιλήσατε για ε, εθνική κυριαρχία. Ε, ναι, τα θέματα εσωτερικής ασφάλειας είναι θέματα εθνικά και αυτό το θέμα ε, στην Επιτροπή μας ε, μας απασχολεί και δεν απασχολεί μόνο εμάς αλλά και την κοινή γνώμη γιατί οι ερωτηθέτες στη τελευταία δημοσκόπηση ε, είπαν ότι το μεγαλύτερο μέλημα όλων των Ευρωπαίων είναι η ασφάλεια περισσότερο και από την ανεργία. Ακόμη και στη δική σας χώρα και στη, και στη Γαλλία να μην μιλάμε τώρα για γαλλογαλλικά μόνο φαινόμενα αλλά Με τις εξαιρετικές γνώσεις σας νομίζω μας ε, δείξατε το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε ε, και σίγουρα έχετε γεννήσει πολλές παρατηρήσεις, ε, ερωτήσεις για τους συναδέλφους. Είναι εξαιρετικά σημαντικά αυτά τα ζητήματα και σίγουρα πέρα από την διαλειτουργικότητα Ε, και αυτή την πρόταση που είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Θα υπάρξουν και άλλες ερωτήσεις. Ε, λοιπόν, ας αρχίσουμε από αυτό, επειδή είναι το πιο επίκαιρο ζήτημα. Ο Αχνό Ντανζόν ε, θα πάρει το λόγο, η Άννα Γκόμες. Σημειώνω τώρα ποιος άλλος θέλει το λόγο. Η κυρία Βαλενσιάνο, η αντιπρόεδρός μας. Να απαντήσω τώρα. Κατευθείαν. Ναι, ναι. Ε, στο στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί είπαμε η πρόταση κατατέθηκε στις 12 Δεκεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο στόχος είναι η ενίσχυση ε, της ε, Ένωσης για την ασφάλεια Πρόκειται λοιπόν για δύο νέους κανονισμούς. Ο στόχος είναι να καλυφθεί το, η έλλειψη πληροφοριών ε, από την οποία πάσχουμε. Πώς αυξάνοντας ε, την δυναμικότητα των συστημάτων πληροφοριών ε, της Ευρώπης για την διαχείριση των συνόρων και των μεταναστευτικών ρευμάτων και εξασφαλίζοντας μια καλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων για, ανάμεσα στα νέα συστήματα για τους νοριοφύλακες, για τους αστυνομικούς, για τους τελωνιακούς υπαλλήλου και ούτω καθεξής. Αυτή η πρόταση λοιπόν ο, αντιπρόεδρος Τίμερμαν ο κύριος Αβραμόπουλο ε, αναφέρθηκαν στο πνεύμα αυτή τη πρόταση και ο κύριο Σοφλάιρτη αναφέρθηκε σε αυτό. Είπαν ότι ναι, ε, νομιμοποιείται ο στόχο για να αναβαθμιστεί η κατάσταση τη ασφάλεια ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είδαμε ότι σε κάθε περίπτωση τρομοκρατική ενέργεια σχεδόν συστηματικά υπήρξε αυτό το θέμα τη ανταλλαγή των πληροφοριών ή ανεπαρκών πληροφοριών ή καθυστέρηση στην ανταλλαγή πληροφοριών ή αν είχαμε την τάδε δίνα πληροφορία ή το τάδε φάκελο, ίσως, ίσως θα μπορούσαμε να έχουμε συλλάβει κάποιους προτού περάσουν στις πράξεις. Ε, είναι εύστοχες ε, όλες αυτές οι παρατηρήσεις ε, και άρα νομιμοποιείται αυτός ο στόχος. Λοιπόν, ε, συμφωνώ με την, τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, με τον κύριο Φλάγκριτη και με τον ε, ε Αρχή Προστασία των Προσωπικών Δομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επίσης τοποθετήθηκαν ε, στα πλαίσια της ομάδας εργασίας εμπρογνωμόνων που πραγματεύτηκαν αυτό το ζήτημα. Παρότι ο κύριος Φλάιρτη τοποθετήθηκε πρώτα ο, ε, των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και η αρχή προστασίας ε, των προσωπικών δεδομένων έχουν ήδη κάνει μια προκατακτική τοποθέτηση. Και υπάρχει μία ανησυχία, δηλαδή... Ορισμένες φορές Κάποιοι ε, κατασταλτικές ε, δυνάμει, ε, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών διαχείρισης μετανάστευσης, οι τελωνιακοί υπάλληλοι έχουν όλοι διαφορετικούς στόχους και διαφορετικές αποστολές και δυστυχώς έχουν πρόσβαση σε δεδομένα που δεν έχουν σχέση με αυτήν την εντολή τους. Λοιπόν, ε, ποιο κίνδυνο ελοχεύει να υπάρξει ένα, ε, μια σύγχυση ανάμεσα στην επικινδυνότητα και ε, την ε, τρομοκρατία και ανάμεσα σε αυτού που ετούνται άσυλο και των μεταναστών. Από την άλλη και το είπε και ο κύριος Έτσι, μπορεί να πληγούν ε, οι ετούντες άσυλο ή οι μετανάστες. Και ξέρετε, ο περασπιστής των δικαιωμάτων στη Γαλλία ή και σε άλλες χώρες ε, που προσπαθούν να προστατεύσουν τους ε, αλλοδαπούς προέλευσης που διαμένουν στη χώρα ή τους μετανάστες που μετικούν στις χώρες μας. Και λοιπόν, ο Ευρωπαϊκός ελεγκτής είπε τα κράτη-μέλη ε, συγχέουν τους στόχους ασφαλείας και τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και ε, φοβάται ότι για την καταπολέμηση της νομοθεσίας και διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων χρησιμοποιούνται μέτρα ε, χωρίς καμία διάκριση και ο κίνδυνος είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας ε, πλέον να μην διαφοροποιείται από τη διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων και έτσι η αλλοδαπή μπορεί να συγχέονται με τους τρομοκράτες. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Ο, ο επόπτης των δεδομένων εξέφρασε αυτή την ανησυχία και ε, ισχυρίζεται θεωρείται ότι ο μόνος τρόπος να αντιμετωπιστεί αποτραπεί αυτός ο κίνδυνος είναι να ε, καταλήξουμε σε ένα πολύ αυστηρό ορισμό ούτω ώστε να χορηγείται πρόσβαση η απαραίτητη ε, για κάθε ε, σκοπό πρόσβαση και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, ε, αυτός ο στόχος διατηρητικότητας των συστημάτων ε, ε, θα πρέπει να σχεδιαστεί και έχοντας κατά νου την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών και υπευθυμίζω γιατί ψηφίσαμε και τώρα σε εθνικό επίπεδο εφαρμόζουμε ένα νέο κανονισμό ε, είναι η αρχή της νομιμότητας, ε, δηλαδή ε, ξεκάθαρος ορισμός του στόχου διακράτηση των δεδομένων και αρχή της νομιμότητας, αρχή της αναλογικότητας. Λοιπόν, θα πρέπει αυτό το σύστημα να παράσχει συγκεκριμένα χέρια δεν θα τα παριθμίσω τώρα. το μας απασχόλησε και μας και ο Ευρωπαϊκός Ελεγκτής έχει τοποθετηθεί για αυτό το ζήτημα και υπενθυμίζω και κάτι άλλο που δεν είναι θέμα μόνο υπερασπιστή δικαιωμάτων αλλά αφορά όλους όσους έχουν ε, πολύ διαφορετικέ εμπειρίες σε αυτόν το τομέα και δυστυχώς βλέπουμε στα πρόσφατα περιστατικά ότι όλο αυτό το σύστημα είναι άχρηστο εάν δεν υπάρχει αμοιβαία ε, εμπιστοσύνη ανάμεσα στις υπηρεσίες πληροφοριών. Και αν ε, αυτές οι υπηρεσίες πληροφοριών δεν κάνουν ε, αυτό που παραπονιούνται πολύ οι άλλοι ότι δεν κάνουν, δηλαδή ότι δεν τους δίνονται σε σωστές πληροφορίες σε το χρόνο και με διαδοχικό τρόπο. Δηλαδή, το θέμα είναι ε, νομικό, είναι θέμα νομιμοποίησης, ε, ε, αλλά εγκυμονεί πάρα πολλούς κινδύνους και πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε και νομίζω ο κύριος Ντανζόν θα έχει πολλά περισσότερα να πει, πολύ περισσότερα από ότι εγώ. Για το ίδιο θέμα θέλει και ο κύριος Ντεπρέ, οπότε μήπως αν συμφωνείτε να δώσω το λόγο στον κύριο Ντεπρέ πρώτα μια που είναι για τη διαλειτουργικότητα. Και μετά ο κύριος Δανζό Ζεράρ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Είναι πιο πολύ διαδικαστικό για την διαλειτουργικότητα. Συμφωνώ απόλυτα και συμμερίζομαι 100% την ανησυχία του κύριου Τυπού όσον αφορά τις κόκκινες γραμμές ανάμεσα στην προστασία και τα δικαιώματα. Αλλά υπάρχουν κάποια άλλα θέματα που απασχολούν για την διαλειτουργικότητα αν μεθαύριο θα μπορούσαν όλες οι αρχές να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες. Μα έτσι όπως προβλέπεται η διάταξη σήμερα από την Κομισιόν, περιορίζει την πρόσβαση των διαφόρων αρχών στις διάφορες βάσεις δεδομένων και πληροφοριών που έχουμε μέχρι σήμερα. Οπότε το να λέτε ότι δεν ισχύει, δεν ισχύει. Δεν είναι αυτή η διαλειτουργική πραγματικότητα σήμερα. Δεύτερον, θέλω κύριε Τουμπό να μου το αποδείξετε ότι στο κείμενο αυτό για την διαλειτουργικότητα. Το θέμα της ε, μετανάστευσης με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας συνδέεται. Τρίτον, για τα δεδομένα. Δεν υπάρχουν νέα δεδομένα φάση του κειμένου για τη διαλειτουργικότητα. Πρόκειται για τη σύνδεση των παλιών. Η βελτίωση ποιότητας κλπ. δεν προβλέπεται από την διαλειτουργικότητα, αλλά από τα διάφορα κείμενα τα οποία διέπουν τη δημιουργία των βάσεων δεδομένων. Λοιπόν, δεν ξέρω το κείμενό σα ποιο σας το συνέταξε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να του πείτε ότι καλά θα έκανε να ξαναδιαβάσει την πρόταση της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Να απαντήσω. Ο κύριο Δημήτρης Αβραμόπουλο, κύριε Τεπρέ, συμφωνείτε μαζί μου έτσι, είναι υπεύθυνο για την μετανάστευση, για τα εσωτερικά ζητήματα και την Ιθαγένεια και δήλωσε ότι σήμερα βρισκόμαστε στο τελευταίο και το πιο σημαντικό τμήμα των εργασιών μας που έχει να κάνει με την κάλυψη των κενών και την ε, άμπλυνση των γονείων όσον αφορά τη διαχείριση των συνόρων και μετανάστευση. Οι συνοριοφύλακε και οι διάφορε αστυνομικοί και άλλε αρμόδιε αρχέ θα έχουν στη διάθεσή του τι κατάλληλε πληροφορίε για να φέρουν σε πέρα στην αποστολή του. Πρόκειται για ένα εμβληματικό στοιχείο τη πολιτική μα κλπ. κλπ, κλπ. Δεν είναι μετανάστευση αυτό. Λέει ότι πρέπει να έχουν τις κατάλληλες πληροφορίες, αλλά δεν λέει ότι είναι οι ίδιες που θα έχουν και πράγματι και υπάρχουν διατάξεις για την διαλειτουργικότητα που θα διατίθενται στους συνοριοφύλακες και άλλες που θα διατίθονται στην αστυνομία. Ο κύριο Τιμπό, μα το κείμενο της Επιτροπής Ανακοινωθένε τύπου το Δεκεμβρίου λέει το σύστημα πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πληροφορίε παραμένουν κατακριματισμένε στα διάφορα συστήματα. Κάτι το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η χρήση του και κινδυνεύουν έτσι οι πληροφορίες να μα ξεφύγουν για την αντιμετώπιση τρομοκρατία κλπ. Οι σημερινές προτάσεις θα καλύψουν τα κενά αυτά και θα φροντίσουν οι πληροφορίες που δίνονται στους συνοριοφύλακες και την αστυνομία να είναι πλήρης και ακριβής. Αφού λέει ότι ο κίνδυνος είναι ο κατακαιρματισμός και ότι αυτό θα διορθωθεί, άρα πάβει να υπάρχει ο κατακαιρματισμός. Δεν το λέω εγώ. Ορίστε, 12 Δεκεμβρίου να κοινωθάνει τίποτα κομισιόν που τα λέει. Ζεράρ, κοιτάξτε. Φυσικά, εγώ που είμαι συνήγορος δικαιωμάτων. Το λέω αυτό και επιμένω. Και όταν μιλάω με βουλευτές, με αρχές και τα λοιπά, με οργανώσεις, συνομιλώ, ανταλλάζω απόψεις και βασίζομαι σε αυτά που μου λένε οι συνομιλητές μου. Συγκεκριμένα εδώ, εσείς και η δική σας επιτροπή. Αλλά, κύριε Ντεπρέ, Λέμε τα πράγματα έτσι ως έχουν και όχι όπως το κάνατε εσείς που με κατηγορείτε ότι εγώ έχω αλλάξει τα δεδομένα. Πρόκειται για ανακοινωθέν Στρασβούργο 12 Δεκεμβρίου 2017. Και τα λέει ξεκάθαρα. Και το πλαίσιο του κειμένου, παρακολουθώντας ε, τις δημόσιες εργασίες των εμπειρογνωμόνων, ακριβώς εκεί καταλήγουν. Γιατί κύριε Ντεπρέ, και πάλι, αν δεν καταλήγαμε στο αποτέλεσμα που λέτε εσείς ότι κατάγειλα και σύμφωνα με εσά δεν υπάρχει, ε, τότε προς τι όλα αυτά. Πρόεδρος. Ε, εκτός μικροφώνου, κύριος Δεπρέ. Επιβεβαιώνω ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν υπάρχουν νέα δεδομένα. Η διαλειτουργικότητα αφορά ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Και δεύτερον, η πρόσβαση στις διάφορες πληροφορίες είναι αυτές που υπάρχουν σήμερα με τις βάσεις δεδομένων που οδήγησαν στα διάφορα συστήματα πληροφοριών. Πρόεδρος. Είναι αλήθεια ότι το θέμα αυτό της αντιπαράθεσης, της πρότασης της Επιτροπής με την διαλειτουργικότητα και οι στόχοι της ε, ασφάλειας για τους Ευρωπαίους είναι θέματα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, τη σημερινή. Ήδη ρωτήσαμε σχετικά τον διευθυντή της ΦΡΑ, θέσαμε τα ρωτήματα και εδώ τώρα στο κύριο Τιμπό. Η συζήτηση που γίνεται σήμερα δείχνει, αν μη τι άλλο, ότι πρέπει να βλέπουμε ξεκάθαρα να ψάξουμε και το άρθρο του Julian King, το χθεσινό, που εξηγείται περί διαλειτουργικότητας. Και σίγουρα θα δουλέψουμε πάνω σε αυτό όλοι. Αλλά δεν πρέπει να καταλήξουμε σε ένα πινκ-πονγκ ε, τυμπον και ενό μόνο συναδέρφου, ο κύριο τυμπον. Βέβαια, αυτό που είναι αλήθεια, λέει ο κύριο τυμπον, είναι ότι στην πρόταση, στην ανακοίνωση της Κομισιόν και λοιπά, δεν πρόκειται για νέα δεδομένα. Πρόκειται για αυτό που ονομάζουν μεγιστοποίηση του ωφέλους από τις πληροφορίες που έχουμε. Αλλά στη σελίδα 2 του εκκαινοθέντων λέει όταν εξηγούμε ότι θέλουμε να αποφύγουμε τις πολλαπλές ταυτότητες, τι σημαίνει αυτό. Ο κύριος Ντανζόν τώρα. Αρνό Ντανζόν για την ερώτησή του. Παρακαλώ. Η ερώτησή μου δεν έχει να κάνει με αυτά μεν, αλλά εποφελούμε για να πω το εξή. Προσοχή, όταν μιλάμε να μην υπάρχει κατακαιρματισμός δεν σημαίνει συγχώνευση. Υπάρχουν διαδικασίες, θα δημιουργηθούν δηλαδή πασαρέλες. Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι θα περνάνε από αυτές τις πασαρέλες, οπότε προσοχή τι γλώσσα χρησιμοποιούμε, τι ορολογία χρησιμοποιούμε. Δεν σημαίνει ότι όλοι θα έχουν πρόσβαση σε όλα. Λέει ότι από αυτά που υπάρχουν σήμερα θα παραμένει διάκριση, δεν θα μπουν όλα μαζί σε ένα καλάθι. Προσοχή. Τώρα, αγαπητέ Ζακ ευχαριστώ που ήρθατε και για την παρουσίασή σας. Εγώ δεν είμαι από αυτούς τους ιστερικούς υπέρ της προστασίας, ακόμα και μεταξύ της δικιάς μου πολιτικής οικογένειας και θέλω να αποφύγω κάθε δημαγωγία που έχουμε κάθε τόσο και μετά τα τραγικά γεγονότα στη Γαλλία που επενθύμησες. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολος είναι ο ρόλος των εσωτερικών για να αποφεύγονται υπερβολές και η υπερβολική ε, νομοθέτηση, ο πληθωρισμός στην νομοθεσία. Το πιο καλό είναι η καλή οργάνωση. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτά. Συμφωνώ. Εκεί όμως που είμαι πιο επικριτικός σε αυτά που ακούω είναι για το ότι η νομοθεσία στη Γαλλία τόνισε πολύ περισσότερο την ασφάλεια σε σχέση με την προστασία των ελευθεριών. Εδώ νομίζω ότι υπάρχει μια αναστροφή της υπόνοιας στη Γαλλία. Δηλαδή, με αυτό θέλω να πω ότι προφανώς κάθε διάταξη, κάθε νομοθεσία, η οποία εξάλλου προσωρινά έτσι, ενισχύει μια διοικητική αρχή, προφανώς και γίνεται σε βάρος του δικαίου και του κράτους δικαίου. Το κράτος δικαίου της Γαλλίας βασίζεται στην διοικητική δικαιοσύνη, έτσι, μεταξύ άλλων, που έχει λόγο ύπαρξης, που έχει τις δικές της προσφυγές, που δεν είναι ο διαιτητής και μερικές φορές στη Γαλλία έχω την αίσθηση ότι την ε, διοίκηση και την δικαιοδοσία της διοίκησης την ταυτίζουμε με το αυθαίρετο. Για τις διαδικασίες που ξεκίνησαν όσον αφορά τους ύποπτους για τρομοκρατικές ενέργειες, τελικά όλα περνάνε από τη δικαιοσύνη, έτσι. Δεν υπάρχει διοικητική δικαιοσύνη που λειτουργεί στο περιθώριο της πραγματικής δικαιοσύνης, οπότε μπορούμε να μιλάμε για Περιορισμού της ποινική δικαιοσύνης, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο και περιορισμένο και στο χρόνο. Έπειτα, οι διώξει. Και όταν λέμε για τη στέρηση ελευθερία με την κράτηση, εγώ δεν συμφωνώ με την ερμηνεία που έγινε, που λέει ότι ο συνήγορο δικαιωμάτων συστηματικά θα πρέπει να αντιτίθεται στις διώξεις και τα λοιπά, γιατί θα σας κατηγορήσουν αν αμέσως δεν κάνετε κάτι. Εγώ έχω παραδείγματα από την προηγούμενη εβδομάδα στη δικιά μου την περιφέρεια, όπου εκεί οι αρχές ακριβώς πέρασαν από το Ζίλντε ζητώντας διώξεις και τους τις αρνήθηκαν. Και τους το αρνήθηκαν και επιπλέον ο υπεύθυνο για τις ελευθερίες σήμερα προηγείται Μερικές φορές βέβαια κάνουμε τα πράγματα ανάποδα. Δηλαδή, δεν είναι αφαίρετο όταν προχωράμε σε κάποια δίωξη, εφόσον υπάρχουν υπόνοιες που πρέπει βέβαια να αιτιολογούνται, αλλά ένα αίτημα ε, έρευνας στο σπίτι κάποιου και δίωξης. Προσοχή μην καταλήξουμε και στον άποδο, να μην μπορούμε δηλαδή να προβούμε στην έρευνα αυτή. Τώρα, για τις προσφυγές που γίνονται. Υπάρχουν 110 περιπτώσεις τα τελευταία δύο χρόνια στον συνήγορο δικαιωμάτων, έτσι. Εγώ δεν νομίζω ότι εδώ παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, γιατί υπενθυμίζω ότι οι άνθρωποι αυτοί στους φακέλους οι οποίοι, για τους οποίους υπάρχουν υπόνοιες πλαστικοποίησης είναι 12.000. Η υπηρεσία πληροφοριών λοιπόν και η Γαλλική Αστυνομία δουλεύει πάνω σε 12.000 άτομα που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί. Ναι, πρόκειται για τους φακέλους ριζοσπαστικοποίησης. Είναι το FSPRT. Εγώ δεν μιλάω για τους φακέλους S, γιατί ξέρω ότι αυτοί δεν απασχολούν τις υπηρεσίες πληροφοριών. Όχι. Οι άνθρωποι που παρακολουθούνται λοιπόν είναι άτομα τα οποία έχουν, για τα οποία έχουν υπάρξει υπόνοιες ριζοσπαστικοποίησης και έχουν σημανθεί έτσι ως ριζοσπαστικομένοι. 12.000 περιπτώσεις, ενώ 110 έφτασαν στο συνήγορο δικαιωμάτων. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι σκανδαλώδες όσον αφορά την αναλογικότητα. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό, ότι ό,τι επικρίσεις και αν μπορεί υπάρχουν και φυσικά και ο συνήγορος δικαιωμάτων πρέπει να κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν νομίζω ότι εδώ έχουμε πλήξει υπερβολικά τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Και ακόμα για μένα, γιατί υπάρχει αυτή η υπόνοια συστηματικά για το γεγονό ότι μια διοικητική αρχή προσωρινά μεν, αλλά στα πλαίσια πάντα του νόμου επίσης, θεωρείται ύποπτη για αυθαιρεσίες. Και μόνο το δικαστικό σώμα, πέρα από το άρθρο 166 του συντάγματος, μπορεί να επιτρέψει τον έλεγχο και την καλή λειτουργία όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι ερωτήσεις του κύριου Νταζά είναι σε πολύ βασικά πλαίσια και απαντώ ως εξής. Πρώτον, δεν υπάρχει καθόλου ιδέα ότι η διοικητική αρχή εξορισμού είναι αφαίρετη ή υδρά κάνοντας διακρίσεις. Όπως το και ο κ. Νταζάν, είναι το άρθρο 166 του συντάγματος που καθιστά τον δικαστή υπεύθυνο για την προστασία των ελευθεριών. Αλλά εδώ και δεκαετίες ο διοικητικός δικαστής έχει αναγνωριστεί στην πραγματικότητα ως αυτός που προστατεύει και τις ατομικές ελευθερίες και τις ελευθερίες γενικά. Υπάρχει απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου και είναι ξεκάθαρο αυτό. Εξάλλου, πρόκειται για μια καινοτομία του καθεστώτος έκτακτης ανάγκης του 2015 που η που πρόθεσε, κάτι που το οποίο δεν υπήρχε στην νομοθεσία του 1955, τη δυνατότητα να υποβάλλεται στον έλεγχο του διοικητικού δικαστή μέτρα έκτακτης ανάγκης, όπως αποφάσεις για έρευνες κατοίκων. Όμως ο διοικητικός δικαστής, ακόμα και στις διαδικασίες αυτές τις έκτακτες, λογοδοτεί αποστεριόρι, δηλαδή είναι υπεύθυνο για την νομιμότητα του μέτρου, είναι υπεύθυνο και απέναντι στην αρχή που πήρε την απόφαση και είναι πάντα υπεύθυνο και λογοδοτή αφού έχει λάβει χώρα και ενέργεια και η πρόοδος της νομοθεσίας της 30ης Οκτωβρίου μετά από αίτημα της ε, νέας πλειοψηφίας μετά τις εκλογές του Ιουνίου είναι ακριβώς η εισαγωγή του ΖΕΛΔΕ και η πλειοψηφία ε, στην ε, Γαλλική Συνέλευση και στη Γερουσία που δεν είναι ίδια συμφώνησαν για την εισαγωγή του ΖΕΛΔΕ. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική προστασία είναι ο απριόρι έλεγχος ενός ε, δικαστή σε σχέση με τον έλεγχο ενός διοικητικού δικαστή ο οποίος αναγνωρίζεται απόλυτα ότι είναι υπεύθυνο για την προστασία του, των ελευθεριών αλλά αυτό γίνεται αποστεριόρι. Και προσθέτω εδώ ότι στην πραγματικότητα 4.500 μέτρα ελήφθησαν από την αρχή της ε, κατάστασης εκτακτής ανάγκης. Και αν υπάρχουν 110 προσφύγες, υπήρξαν χίλιες δικητικές περιπτώσεις ακριβώς. Οι περισσότεροι είχαν την τάση να πούν θα απευθυνθώ στο δικητικό δικαστήριο θα υποβάλω αίτημα στο στεγματικό δικαστήριο, ξέρω τι, αντί να έρθει να δει τον ε, συνήγορο δικαιωμάτων, που υπενθυμίζω ότι η αρμοδιότητά του εξαρτάται από την διοντολογία που διέπει την ασφάλεια. Καθορίζεται στον κώδικα εσωτερικής ασφάλειας. Επίσης, έχω και την εξή παρατήρηση για αυτά που είπε ο κ. Ντανζό. Ακριβώς μετά από όλα τα διοικητικά μέτρα που ελήφθησαν, όντως υπήρξαν ελάχιστες δικαστικές υποθέσεις που προχώρησαν για την τρομοκρατία. Υπήρξαν πολλές δικαστικές υποθέσεις που είχαν να κάνουν με τα ναρκωτικά, όπλα, εγκληματικότητα του κοινού δικαίου. Αλλά πραγματικά μετρώτε στα δάχτυλα του ενός χεριού οι περιπτώσεις που είχαν να κάνουν με την τρομοκρατία που πέρασαν από αυτές τις διοικητικές διαδικασίες. Και στην πραγματικότητα το βασικό που έγινε και βοήθησε να αποφύγουμε τρομοκρατικές ενέργειες, να αποτελεσματικοί δηλαδή στην πρόληψή τους, αυτό έγινε μεταξύ έργου υπηρεσιών πληροφοριών εκτός χώρας, εντός της χώρας, που στη συνέχεια πήγαν στο αντιτρομοκρατικό σώμα, το οποίο έδρασε έγκαιρα. Δηλαδή είναι ο καλύτερος τρόπος για την πρόληψη. Και αυτό συνδέεται και με αυτό που είπαμε πριν. Γιατί να τα κάνουμε όλα αυτά αλλιώς. Αλλά δέχομαι βεβαίως αυτό που είπες ότι το GLD πρέπει να είναι αποτελεσματικό. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε πολύ για την απάντηση αυτή. Η κυρία Αναγκόμες. Ευχαριστώ κύριε Τουμπό για όλα αυτά που μας είπατε, πολύ ενδιαφέροντα. Μιλήσατε για μέτρα τα οποία δοκιμάστηκαν στη Γαλλία όσον αφορά τα άτομα που έχουν δύο επικότητες, κάτι το οποίο κατέληξε στην παρέτηση της κυρίας ε, Τομπίρα, είναι προς τιμή της. Η κυρία Στίβενς που είναι η συνηγήτρια δεν είναι εδώ, αλλά πριν ρώτησε κάτι τον κύριο Φλάερτη για τις εκδόσεις υπόπτων. Και θέλω να σας ρωτήσω, με τη συζήτηση που έχετε κάνει στη Γαλλία από αυτόν, και με όλα όσα γνωρίζετε εσείς. Η ιδέα αυτή τρελή κατά τη γνώμη μου. Να εκδίδουμε υπόπτους. Διασφαλίζει τον έλεγχο των υπόπτων αυτών πιο αποτελεσματικά. Από ότι αν θα μπορούσαμε να τους κρατήσουμε στη Γαλλία, έτσι όπως μας τα έχετε περιγράψει ότι ισχύουν εκεί. Δηλαδή, σε μια χώρα όπως είναι το Μαρόκο ας πούμε, γιατί πολλοί υποπτοί προέρχονται από το Μαρόκο. Θα μπορούσαμε στο Μαρόκο δηλαδή να περιμένουμε ότι εκεί η δικαιοσύνη θα τους αντιμετώπιζε αποτελεσματικά. Και δεν μιλάω μόνο για την ασφάλεια εδώ, μιλάω και για τις ε, δίκες. Αν δηλαδή όντως οι άνθρωποι αυτοί μπορούν να αποδειχτούν τρομοκράτες σωστά. Απάντηση του κύριου Τιμπού. Στο κράτος δικαίου έχουμε πάντα μέτρα τα οποία επιτρέπουν να απομακρύνουμε από τη Γαλλία, να εκδίδουμε άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί. Υπάρχει τέτοια διαδικασία. Δεν αφορά τα άτομα τα οποία είναι ύποπτα ότι έχουν κάνει το ένα ή το άλλο. Δεύτερον, όσον αφορά τα μέτρα που θα μας επέτρεπαν την έκδοση των ατόμων αυτών, των υπόπτων αυτών, πράγματι στη δημόσια συζήτηση διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν άτομα, κόμματα και λοιπά που έχουν κάνει τέτοιες προτάσεις. Αλλά ειλικρινά εγώ έχω την αίσθηση, θα με λέξει εδώ και ο κύριος Ντονζό, ότι ποτέ δεν πήγαμε μακριά από αυτού. Και το μόνο ζήτημα που ετέθη είναι το θέμα των ατόμων που έχουν διπλή υπηκότητα πράγματι, αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γιατί αυτό σημαίνει ότι τελικά δεν είναι η γαλλική υπηκότητα όταν έχουν καταδικαστεί, έτσι. Αφόσον λοιπόν δεν έχουν την γαλλική υπηκότητα, μπορούμε να θεωρήσουμε, μπορούμε και να τους διώξουμε. Τέλος. Παρά τη σοβαρότητα του θέματος, που είναι τραγικό, μπορώ να σας πω με ένα χαμόγελο, ότι διαπιστώσαμε ότι αυτό που κάνει καλύτερα ο τρομοκράτης είναι να κατέχει πολύ καλά τι μπορεί να κάνει στο τρένο, στο αεροδρόμιο, με το αεροπλάνο, στους σταθμούς κτλ. Δηλαδή το να νομίζουμε ότι επειδή τους διώξαμε δεν θα ξανάρθουν είναι ψευδέστηση. Εφόσον δεν έχουμε διασφαλίσει μια πολύ καλή εποπτεία και παρακολούθηση. Έτσι, αυτό είναι πάντα το ζήτημα. Για το Μαρόκο δεν θέλω να εκφραστώ, αλλά για να είμαστε αποτελεσματικοί θα έπρεπε τα άτομα αυτά να τα στέλνουμε σε χώρες όπου είμαστε σίγουροι ότι θα έχουν μια αντιμετώπιση που να συνάδει απόλυτα με τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Καταλαβαίνω ότι δεν βρισκόμαστε εκεί. Αλλά η πολιτική ασύλου και μετανάστευσης μπερδεύεται πολλές φορές. Όμως υπάρχουν μέτρα σε αυτή την περίπτωση για το άσλολο και τους μετανάστες βάσει των οποίων στέλνουμε τους ανθρώπους αυτούς σε χώρες που θεωρούμε ασφαλείς ενώ δεν είναι καθόλου ασφαλείς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είναι σίγουρες αυτές οι χώρες, δεν είναι ασφαλείς. Μάλιστα, παράκαμψη ήταν αυτή. Εντάξει, αλλά ξεκάθαρη η γλώσσα σας. Μα θα τεθεί το ερώτημα. Γιατί το Συμβούλιο και η Κομισιόν συζητούν αυτή την εποχή τον κανονισμό που έχει να κάνει με τις τρίτες ασφαλείς χώρες. Πρόεδρος, ναι, είναι ζωτική σημασία σε αυτό και είναι ένα θέμα όμως που σέρνουμε εδώ και πολύ καιρό με τις συμφωνίες επανεισδοχής με το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, πώς οργανωνόμαστε. Ο δρόμος είναι μακρύς, ε. Τι κάποιος έλεγε τις προάλλες πριν από δεκαετίες είχε συζητηθεί η σύμβαση της Γενέβης και φαίνεται ότι ήδη τότε είχε τεθεί το θέμα του ποιες χώρες θεωρούνται ασφαλείς και ποιες όχι. Πρόεδρος, ευχαριστούμε η Έλενα Βαλενθιάνο τώρα, που είναι αντιπρόεδρος στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ, θα μιλήσω ισπανικά, για να μην έχουμε γαλλική συζήτηση μόνο. Τι να κάνουμε. Ευχαριστούμε που ήρθατε να συζητήσουμε για αυτά τα θέματα και διαπιστώνουμε ότι όντω υπάρχει μια ανισορροπία υπέρ τη ασφάλεια και σε βάρο των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, δεν το συζητάμε υποθετικά, το ξέρουμε ότι συμβαίνει. Έτσι. Θέλαμε ισορροπία, αλλά δεν υπάρχει ισορροπία. Εδώ και καιρό το λέμε. Και τελικά έχει κερδίσει ασφάλεια σε βάρος των δικαιωμάτων επειδή η κοινωνία το ζητά, επειδή η κοινωνία εκφράζει όλο και μεγαλύτερη ανησυχία για την ασφαλειά της. Αλλά και για την ελευθερία της. Τέλος πάντων, φοβάται η κοινωνία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οπότε, το να νομοθετούμε βάση μιας τραυματικής εμπειρίας δεν μας οδηγεί πουθενά. Γιατί όλο και νέα τραύματα θα έχουμε και όλο και θα σκληραίνει η νομοθεσία και η ασφάλεια θα υπερισχύει κάθε φορά όλο και περισσότερο. Θεωρείται εντελώς κανονικό πια ζήτημα ο έλεγχος στα αεροδρόμια. Ναι, αλλά έχει αξιολογήσει κανείς, έχει εκτιμήσει πόσο κοστίζει αυτό το σύστημα ελέγχου σε σχέση με τις επιθέσεις που έχουμε αποφύγει στα αεροπλάνα. Έχει διαπιστώσει κανείς τη σχέση αυτών των συστημάτων που είναι υπερβολικά και που δυσκολεύουν πάρα πολύ τη ζωή πολλών Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων, κυρίως των μη Ευρωπαίων. Εξυπηρετούν αυτά τα συστήματα για να πετύχουμε τον στόχο μας. Αυτό είναι το ζήτημα. Αν δηλαδή συστηματικά προσπαθούμε να πετύχουμε την ισορροπία, μήπως θα έπρεπε να ε, μετρήσουμε και τη ζημιά εντό εισαγωγικών που έχει γίνει στους ανθρώπους που έχουν ε, δυσκολευτεί, που έχουν ταλαιπωρηθεί από όλα αυτά τα συστήματα και να το βάλουμε αυτό στη ζυγαριά με αυτά που έχουμε πετύχει. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ντυπό. Θα έλεγα ότι γενικά μιλώντας τα μέτρα που λαμβάνονται πρέπει να λαμβάνονται εκτός βέβαια αν εμπλέκεται το συνέστημα ε, θα έπρεπε λοιπόν να λαμβάνονται αλλά ορθολογικά πιο ορθολογικά και αυτό είναι το ζήτημα το δίκαιο μας δίνει απαντήσεις που βασίζονται σε επιχειρηματολογία που αυτή βασίζεται στις αρχές μας, στις θεμελιώδεις αρχές μας και που είναι απόλυτες. Οπότε μερικές φορές απέναντι σε αυτά υπάρχουν άλλα πράγματα που δεν είναι ορθολογικά που υπερισχύουν. Συχνά μάλιστα για τα μέσα ενημέρωσης και από εκεί και πέρα αναγκαζόμαστε να κάνουμε πράγματα. Να, για παράδειγμα, πριν από δύο χρόνια υπήρξε ένας πολύ σημαντικός υπεύθυνο των υπηρεσιών πληροφοριών σε μια επιτροπή, δεν ξέρω τώρα αν της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης ή της Γερουσίας, που είπε, αν θέλετε να σας πω πραγματικά τι πιστεύω, τα μέτρα αυτά λαμβάνονται για να καθισχαστεί η κοινή γνώμη. Ότι δηλαδή πράγματι η κυβέρνηση κάνει κάτι, δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια. Εντάξει, τώρα εννοείται ότι αυτό που έλεγε ο άνθρωπος ήταν ότι αν μου δίνατε περισσότερα μέσα εγώ θα έκανα πιο αποτελεσματικά πράγματα. Και είχε δίκιο. Έτσι. Αλλά τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται και αυτό το εμείς καταγγείλαμε στο σχέδιο νόμου για τις πληροφορίες, ότι τα μέτρα δεν πρέπει τελικά να θέτουν υποφυσβήτηση τις λεθερίες να είναι τόσο δηλαδή παρεμβατικά που να περιορίζονται αυτές. Αυτό που είπατε για την ασφάλεια των αεροπλάνων είναι ακριβώς χαρακτηριστική επιχειρηματολογία. Φανταστείτε μεθαύριο εδώ που βρισκόμαστε τώρα, έτσι. Φτάνετε σε ένα αεροδρόμιο και φτάνετε στην είσοδο του αεροπλάνου χωρίς να σας συζητήσει κανείς τίποτα. Εσείς, τόσο πάντων όχι εσείς, αλλά οι άλλοι τι θα σκεφτούν, θα σκεφτούν με τρελάθηκαν, δεν ελέγχεται πια κανείς. Όποιο να είναι μπορεί να μπει σε αυτό το αεροπλάνο χωρί έλεγχο, μα θα το ανατινάξει. Βρισκόμαστε δηλαδή σε μια κατάσταση, σε ένα κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία μας. Τέτοιο που απαιτεί τα μέτρα. Λοιπόν, είπα, πρέπει να λαμβάνονται με ορθολογικό τρόπο. Συμφωνώ. Και κύριε Νταζά, κάτι ακόμα νομίζω ότι αυτό θέλατε να πείτε πριν. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα διάταξη στη, στο νομοθεσία της 30 Οκτωβρίου λέει ότι δεν θα εφαρμοστεί παρά μέχρι το 2020 και ότι τότε το 2020 θα εκπέσει. Και τότε θα συζητήσουμε αν οι διατάξεις που έχουν ληφθεί τελικά ήταν αποτελεσματικές ή όχι, άρα αν πρέπει να τις διατηρήσουμε, αν πρέπει να εξαφανιστούν ή να τροποποιηθούν. Είναι λίγο πολύ αυτό που είπατε κι εσείς. Φυσικά κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η κατάσταση της χώρας και της Ευρώπης και της κοινή γνώμης το 2020. Όμως είναι μια προσπάθεια που πάει προς την κατεύθυνση αυτό που είπατε και εσείς κύριε Αντιπρόεδρε. Ζακ Τουμπό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, έχετε το λόγο αν θέλετε. Έχουμε ακόμη λίγο χρόνο αν ε, έχετε άλλες ερωτήσεις. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Ακόμη δεν μιλήσαμε για τη δημόσια γνώμη, για το σοκ της δημόσιας γνώμης και χθε ε, που ήταν ε, που θυμηθήκαμε όλη αυτή τη βάρβαρη τρομοκρατική ενέργεια που οδήγησε σε τόσα πολλά θύματα στις χώρες μας ε, και βήθησε στο πένθος τη Γαλλία, τίποτα ε, δεν επέστρεψε στη κανονική κατάσταση μετά τον Ιανουάριο του 2015. Και ε, δίκαιο έχετε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό γιατί και εγώ νομικός είμαι και συμφωνώ. Ε, και μην ξεχνάμε ότι αποτρέπονται ε, τρομοκρατικές επιθέσεις καθημερινά στη Γαλλία και επειδή μιλήσαμε και για άλλες χώρες ζητώ συγγνώμη για τους συναδέλφους ε, ε, στη σημερινή συνεδρία ήταν γαλλικά όλα τα παραδείγματα που δώσαμε. Υπάρχουν όλα και περισσότερα εργαλεία αντιτρομοκρατικά και Υπάρχουν και κάποιοι που ισχυρίζονται ότι ε, και τίποτα να μην κάναμε το ίδιο θα ήταν το αποτέλεσμα. Εγώ αντίθετα πιστεύω ότι υπάρχουν πολύ χρήσιμα εργαλεία και είναι πολύ ε, σοβαρές οι απειλές ε, κατά της Γαλλίας και αποτρέπονται καθημερινά τρομοκρατικές συνέργειες και γι' αυτό και ε, βρίσκεται σε σοκ η δημόσια γνώμη και θα πρέπει ε, να υπάρξουν αποδείξεις όπως και στην αγάπη ε, δεν μπορούμε απλώς να τους καθησυχάσουμε πρέπει να ε, αποδείξουμε ότι θα κάνουμε αρκετά ούτως ώστε να βγούμε νικητές σε αυτόν τον αγώνα κατά της τρομοκρατίας είναι υπαρκτές οι απειλές, οι φόβοι και όσοι φέρουν τις ευθύνες οφείλουν να ε, ανταποκριθούν ε, στη, στη δημόσια γνώμη γιατί επικρατεί ο φόβος. Ε, Πρόεδρε, πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε, αλλά δυστυχώς δεν αποφασίζω εγώ το πρόγραμμα εργασίας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, σήμερα μα μένει ο κ. Φλάγερτη από τον οργανισμό που φυσικά δεν είναι αποκομμένο από την εκτελεστική εξουσία, αλλά ε, μα μίλησε για το ζήτημα των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είναι ε, πάρα πολύ ενδιαφέρον το ζήτημα. Αν ακούσετε τι πιστεύουν κάποιες ισπανικές αρχές ε, ή το Συμβούλιο της Επικρατείας, ε, το Σταγματικό Δικαστήριο στην Καλσούη ή ε, οι Αγγλικές Αρχές, θα ακούσετε διαφορετικές απόψεις ανάλογα με τη δική τους ε, ε, ένωμη τάξη. Και τώρα τι, δεν μετράμε αριθμό θυμάτων, ε, γιατί εξάλλου η, προ... ε, τρομοκρατική ενέργεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Γερμανοί είχαν να αντιμετωπίσουν αυτή την επίθεση στη χριστουγεννιάτικη αγορά και όπως και η Ιταλία έχουν άλλα ιστορικά βιώματα ε, η Ρότε Φραξιόν στην ε, Γερμανία οι Ερυθρές Ταξιαρχίες στην Ιταλία υπάρχει δηλαδή ιστορικό βιώμα παράδοση και από τη δεκαετία του 70 έχουμε αποφάσεις ε, του Συνταγματικού Δικαστηρίου που έχουν ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και αυτό το είπα για να μην μου λέτε ότι φέρνω μόνο γαλλικά και βρεξελιώτικα παραδείγματα. Ε, ναι, ε, για να έχουμε και το δικαστήριο της Καστρούης μπορούμε να συναντηθούμε με γερμανικές αρχές και ισπανικές αρχές. Θα δώσω το λόγο στον Αχνό Ντανζό και στην Κατερίνα Κινίτσι. Θέλω να πω στον Ζακ Τουμπό ότι συμφωνώ με δύο πολύ σημαντικά σημεία της ανάλυσης του για την αντιτρομοκρατική δράση. Αυτό που καθησυχάζει δεν ε, ε, είναι κάτι που απαραίτητα προστατεύει. Ε, αυτό αληθεύει για πολλούς έκτακτους μηχανισμούς που έχουν στόχο να καθησυχάσουν, αλλά από πλευράς αποτελεσματικότητας θα πρέπει να αξιολογηθούν ενδελεχέστερα. Επίσης, ε, ο νομικός μηχανισμός, όσο εξελιγμένος, όσο λεπτομερής και αν είναι, μην ξεχνάμε ότι ο αριθμός, ο βαθμός λεπτομέρειας ε, δεν είναι εγγύηση αποτελεσματικότητας. Ε, μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για υπηρεσίες πληροφοριών και κατασταλτικές αρχές που είναι πολύ πιο προηγμένες από αυτή την άποψη. Αλλά τέλος πάντων... Ε, πιστεύω ότι ε, δεν πρέπει να διακομωδούμε γιατί η ανταλλαγή είναι πολύ καλύτερη από όσο ισχυρίζονται πολλοί. Πάλι θα αναφερθώ σε μια γαλλική περίπτωση, αλλά τι να κάνω. Μιλήσαμε για την ειδική την αντιτρομοκρατική ε, εισαγγελία στον, στο παρελθόν. Ο εισαγγελέας Μολά ε, θεωρούσε ότι ήταν ικανοποιητικό το σύστημα που υπήρχε μην ξεχνάμε ε, αριθμητικά και μόνο πόσο ε, πολλοί είναι οι υποθέσεις που πρέπει να διερευνηθούν και ίσως αναπόφευκτα ε, θεσπιστεί ε, μια ανεξάρτητη εισαγγελία, μήπως ε, και πάλι είναι επικοινωνιακή η δράση, δηλαδή να δώσουμε την εντύπωση ότι θα ειδικευτεί η εισαγγελία και θα είναι άρα πιο αποτελεσματική, ενώ μέχρι τούδε η εισαγγελία δεν λειτουργούσε ικανοποιητικά, ενώ αυτό δεν ισχύει απαραίτητα. Ζακ του Ε, φυσικά δεν μιλούσα για την ε, οργάνωση, ε, τη δικαστική οργάνωση και την πολιτική που ακολουθείτε, διότι δεν είναι δική μου αρμοδιότητα και, και δεν είναι και του παράντος, δεν είναι το θέμα μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. εγώ Ήμουν ε, πρόεδρος της Νομοτεχνικής Επιτροπής ε, το 86 όταν θεσπίστηκε η, αυτός ο αντιτρομοκρατικός μηχανισμός στη Γαλλία μετά από τις ε, επιθέσεις του 86. Ε, λοιπόν... Οι δράστες ήταν από τη Μέση Ανατολή τότε. Ο μηχανισμός λειτουργεί εδώ και 30 χρόνια και η ποιότητα του ε, είναι συνάρτηση της αποτελεσματικότητας του, αυτό ανέκαθεν το πρέσβευε και έχετε επίση το σεβασμό των διαδικασιών του ποινικού δικαίου. Δηλαδή δημιουργούνται θύλακες ε, μέσα ε, στην διαδικασία του ποινικού δικαίου, όμως ταυτόχρονα διατηρείται η συνοχή σε σχέση με ολόκληρο τον μηχανισμό του ποινικού δικαίου και άρα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε όπως είπε ο κ. Μαρτή ή όπως ε, συζητήσαμε προηγουμένως δεν πρόκειται για ε, ζήτημα εσωτερικής ασφάλειας, ε, παραμένει ε, αναπόσπαστο κομμάτι του ποινικού δικαίου και συγκεντρώνονται στην εισαγγελία στο Παρίσι όλες οι υποθέσεις εάν υπάρξει συνάφεια. Αυτή η οργάνωση ε, με τρομοκρατικό στόχο, λοιπόν, όταν συστήνεται, δηλαδή με το που χαρακτηρίζεται ε, αυτή η συνάφεια, τότε ε, δρομολογούνται όλες οι υποθέσεις προς την εισαγγελία του στο Παρίσι. Δεν έχω την εντύπωση ότι είναι ατέλης και ότι στερεί αυτός ο μηχανισμός. Έχουν ε, φυσικά αλλάξει οι περιστάσεις, η κατάσταση, αλλά δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι ελαττωματικός αυτός ο μηχανισμός. Επίσης, από τεχνικής πλευράς έχουν την εισαγγελία στο Παρίσι, την ε, εθνική, ε, αυτή η εισαγγελία που προτάθηκε να συσταθεί δηλαδή για τις τρομοκρατικές υποθέσεις Ποια είναι η απόψή μου. αυτό ο μηχανισμός, δηλαδή από τι τοπικέ εισαγγελίε, να πηγαίνουμε στην κεντρική, από τι υπηρεσίε πληροφοριών σε τοπικό επίπεδο να ανεβαίνουμε στην εισαγγελία στο Παρίσι, με το που χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση, δεν είναι αυτό το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου. Οπότε ε, η εναλλακτική λύση που είναι μια δικαστική ε, απόφαση, εάν γίνει, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Η εισαγγελία του Παρίσι δεν θα έχει πλέον αυτές τις τρομοκρατικές υποθέσεις και άρα θα έχει μεγαλύτερη ευχέρεια να επιληφθεί άλλων σημαντικών ε, ζητημάτων για τα οποία φέρει την ευθύνη. Αυτό πιστεύω, Αρνό. Αυτά είναι τα αρχή, αλλά νομίζω ότι θα γίνουν διεξοδικότερες ε, συζητήσεις για αυτό το ζήτημα και ο υπουργό δικαιοσύνη νομίζω τώρα αυτή τη στιγμή ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά ε, ενός τέτοιου μέτρου. Υπάρχουν και παραδείγματα από άλλες χώρες. Υπάρχουν... Υπάρχουν όλα τα πιθανά σενάρια. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να, απλώς να συγκρίνουμε και να λέμε να κάνουμε αυτό ή εκείνο. Έχουμε το ισπανικό σύστημα, έχουμε πάρα πολλά διαφορετικά. Ο εισαγγελέα Μωράνσε ε, δεν ε, ήταν ε, ε, υπέρ αυτής της ε, άποψης η Κατερίνα Κινήση ε, μπορεί να κάνει την ερώτησή της τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τουμπόν για τις ε, προτάσεις, τις σκέψεις του, για την ε, διαφάνεια και την διανοητική ειλικρίνεια με την οποία το έπραξε. Είναι πολύ χρήσιμες και για τη δουλειά βέβαια της Επιτροπής μας όλες αυτές τις σκέψεις. Όταν μιλούμε λοιπόν για δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα, προστασία δικαιωμάτων, θέλω, όπως είπε και η κυρία Κρίσπεκ, να σταθώ με την ερώτησή μου σε ένα άλλο θέμα, ε, να, να μετατοπίσω το επίκεντρο βέβαια πάντα στα δικαιώματα και φυσικά ε, μην αγνοώντας την τραγική επέτειο της επίθεσης στο Σαρλί όπου μετά τα γεγονότα αυτά ε, γενική αίσθηση των πολιτών ότι τα πράγματα άλλαξαν πια, δεν είναι όπως ήταν πριν. Και επειδή έχω και προσωπική αντίστοιχη εμπειρία, ξέρω και εγώ πολύ καλά ότι τίποτα πια δεν είναι όπως ήταν πριν. Ο πατέρας μου πριν από 35 χρόνια δικαστής ε, εκτελέστηκε από τη μαφία με μια βόμβα μαζί με δύο καραμπινιέρους που τον συνδωνεύαν μπροστά από το δικαστικό μεγάλο και πια τίποτε δεν είναι όπως ήταν πριν για τις οικογένειες των θυμάτων και όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να σβήσει κανείς από τα μάτια του και από το η μνήμη του τις εικόνες των τραγικών γεγονότων, αλλά και γιατί ε, είναι όλες οι συνέπειες αυτών των τραγικών γεγονότων παρούσες. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας απασχολήσει, η προστασία και η υποστήριξη των θυμάτων που άλλωστε προβλέπει και η οδηγία. Μίλησαμε λοιπόν για διάφορες πτυχές της προστασίας των δικαιωμάτων ε, των πολιτών, αλλά όχι τόσο των θυμάτων και οικείων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Θα ήθελα λοιπόν τις δικές σας ιδέες για τα όσα έχουμε συμπεριλάβει στην οδηγία, διάφορες μορφές προστασίας που προσπαθήσαμε να εκφράσουμε ως έκκληση προς τα κράτη-μέλη την σχετική προστασία. Πιστεύετε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο, κάτι καλύτερο. Υπάρχουν εμπειρίες από διάφορα κράτη που ενδεχομένω να είναι χρήσιμε ε, για άλλα κράτη. Εκεί όπου υπήρξαν δυστυχώς τέτοιες τραγικές ε, ε, πράξεις. Και σας ευχαριστώ πολύ που αναφέρατε νωρίτερα τη δουλειά που κάναμε μαζί με την πρόεδρο στην Intergroup για τα δικαιώματα των ανηλίκων, γιατί είναι θεμελιωδέστατα τα δικαιώματα αυτά των πιο ευάλωτων εκείνων, των παιδιών που χρειάζονται περισσότερη προστασία και που όπως συμβαίνει συχνά στα περίπτωση των θυμάτων και των οικείων των θυμάτων της τρομοκρατίας του οργανωμένου εγκλήματος αλλά και γενικότερα ε, σε σχέση με τα θύματα ή τους οικείους των θυμάτων ενός αδικήματος, ενός εγκλήματος, έχουμε την εντύπωση ότι είναι λίγο παρόντα σε όλες αυτές τις διαδικασίες ε, και τα όσα προβλέπει η νομοθεσία ή τα μέτρα είναι λίγο παρούσα η προστασία και το μέλημα για ε, τα θύματα και τους οικείους τους. Αλλά ιδιαίτερα σε ευχαριστώ για να ολοκληρώσω για την αναφορά στα δικαιώματα των ανηλίκων και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε βέβαια για να εργαστούμε περισσότερο στο θέμα αυτό. Κύριε Στουμπού. Κυρία Κινίτσι. Πιστεύω ότι όλα αυτά, αν θέλουμε να τα κοιτάξουμε μέσα από το πρίσμα της ιστορίας και βέβαια μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όντας οι αποδέκτες της παρακαταθήκης και του οικοδομήματος της Ευρώπης μετά την τραγωδία του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τη βαρβαρότητα των Ναζί και την τραγωδία της ε, ΣΟΑ. Έχουμε πολλά να πούμε, χωρίς βέβαια να παραμελούμε και τη σημασία, την ιστορική σημασία της πτώσης του τείχους το 89 και της άφηξης όλων αυτών των κρατών έκτοτε, των κρατών εκείνων που είχαν αποστηριθεί τα δικαιώματα και τις εγγύησεις για 40 χρόνια για πολλά από αυτά. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ε, ιστορική προοπτική και το είπατε κι εσείς, όντως τίποτα δεν είναι όπως ήταν πριν. Η 11η Σεπτεμβρίου άλλαξε τα πάντα στις Ηνωμένε Πολιτείες. Δεν είναι τίποτα όπως πριν. Στις Ηνωμένε Πολιτείες αλλά και γενικότερα για οποιονδήποτε με κάποιον τρόπο παρακολουθεί την αντίληψη των Ηνωμένων Πολιτείων σε επίπεδο διπλωματικό, στρατιωτικό, δικαστικό. Είναι σαφές το σύνδρομο της 11 Σεπτεμβρίου σήμερα έχει κατά κάποιο τρόπο εκπεκταθεί σε όλη την Ευρώπη, ύστερα και από τις τρομοκρατικές επιθέσεις του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους και των όσων έλαβαν χώρα στις χώρες μας, τη Γαλλία, τη Γερμανία και άλλες. Τη Δανία, το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ερώτημα λοιπόν σε όρους ιστορικούς είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτό. Θα συνεχίσουμε να λέμε τίποτα πια δεν είναι όπως πριν. Και άρα να εισάγουμε διατάξεις και μέτρα που εξακολουθώ να πιστεύω πως είναι δυσανάλογα σε σχέση με το κράτος δικαίου, αγνώντας όχι το παρελθόν, αλλά αυτό που έχουμε μπροστά μας στο μέλλον. Δηλαδή, το ερώτημα ποιο κράτος δικαίου θα παραδώσουμε στα παιδιά και τα εγγόνια μας. Και σε όσους πολιτικούς θα μιλήσω τώρα, τι κράτος δικαίου θα παραδώσουμε στις μελλοντικέ κυβερνήσεις και τις μελλοντικέ κοινοβουλευτικέ πλειοψηφίες, που ίσως να μην είναι όλες το ίδιο ε, θετικά διακείμενες, να μην σέβονται όλες το ίδιο το κράτος δικαίου και τις αρχές του κράτους δικαίου, είτε στη μια χώρα είτε στην άλλη, είτε παντού. Και αυτό ήταν και ένα από τα μελήματα που ε, τοποθέτησα στο επίκεντρο των ανησυχιών μου. Δηλαδή η κρατική συνοχή, η κοινωνική συνοχή δεν πρέπει να τεθούν σε κίνδυνο με το να στοχεύουμε μέσα στις κοινωνίες μας κάποιους που για διάφορους και σοβαρούς λόγους, το λέμε και στο κείμενο, μπορεί να καταστούν στόχοι της προληπτικής αντιτρομοκρατικής δράσης ως ε, ομάδες κοινωνικές, ως ε, ομάδες θρησκευτικέ, ως ε, άτομα προερχόμενα από μια συγκεκριμένη καταγωγή χώρα. Γιατί αυτό δεν είναι αμεληταίο. Και πάνω απ' όλα πρέπει να φροντίσουμε να μην εισαγάγουμε μέτρα στις ανομές μας τάξεις που αν πέσουν στα χέρια ορισμένων μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τις ελευθερίες. Και εδώ έτσι κυρία Κινίτση επιμένω ότι πρέπει να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα όντω, τίποτε δεν είναι όπω πριν. Βεβαίω και πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη και βέβαια μέσα, αυτή την μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να δράσουμε, αλλά πρέπει και να δράσουμε ε, αναζητώντα το πώ θα ξανασταθούμε στα πόδια μα στο μέλλον και τι θα παραδώσουμε, τι παρακαταθήκη θα αφήσουμε στι μελλοντικέ γενιέ. Και βεβαίω εγώ είμαι μεταξύ εκείνων που πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα απαλληφθεί αυτή η απειλή, κάποια στιγμή θα ξαναβρεθούμε σε μια κατάσταση όπου δεν θα ξυπνάμε κάθε πρωί σκεπτόμενοι ότι μπορεί να εκδηλωθεί μια τρομοκρατική επίθεση μέσα σε ένα λεωφορείο στη γωνία του δρόμου. Με την προπτική λοιπόν αυτή έρχομαι να απαντήσω συναφώς και στη δεύτερη ερώτηση σας. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να μεριμνούμε για τα θέματα, όχι μόνο για να μνημονεύσουμε τις επιθέσεις, τα εγκλήματα, για να εκδηλώσουμε την συμπάθεια και την συνέστησή μας, αλλά να μεριμνήσουμε για τα θέματα ως άτομα και να, τα αντιληφθούμε ως άτομα τα οποία είναι σε θέση από θύματα παθητικά να μεταβούν σε μια κατάσταση άλλη γιατί ναι, μπορεί να αντιμετωπίσουμε καλά τα θύματα, αλλά εάν μπορούν να επανενταχθούν, εάν μπορέσουν να ξαναβρούν με κάθε έννοια προσωπική, επαγγελματική κτλ. μια κανονική ζωή, παρά το τραύμα, παρά το πένθος που έχουν βιώσει και εσείς προσωπικώς μιλήσατε για το δικό σας πένθος, αγαπητή κυρία Κυρίτση. Αν μπορέσουμε λοιπόν αυτό να το κάνουμε, τότε έχουμε φτιάξει μια βάση ανθρώπινη για να περάσουμε σε αυτό το νέο στάδιο το οποίο εγώ εύχομαι να εξασφαλιστεί, δηλαδή να ξεφύγουμε από αυτό που θα ξανααποκαλέσω σύνδρομο της 11 Σεπτεμβρίου, για να μεταβούμε σε ένα άλλο καθεστώ σε μια άλλη κατάσταση και μια και μιλούμε για το δικό μας το κράτος, για την νομοθεσία, τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, την ένωμη μας τάξη. Και έτσι εμείς διατυπώνουμε τις προτάσεις μας, τις ταπεινές αυτές προτάσεις, στο δικό μας το ε, επίπεδο, που όμως ε, εμπνέονται από αυτό το πνεύμα. Και έτσι ολοκληρώνω, μιλώντας πάλι για τη δική μας την το νομίζω ότι ισχύει για τους πάντες... Το καθεστώς αυτό των θυμάτων πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Πρέπει να χτίσουμε αυτή την πρόοδο για τα θύματα χάρη σε ένα ειδικό καθεστώς και μια ειδική μεταχείριση ή πρέπει να ισχύσουν και για τα θύματα τα μέτρα του κοινού δικαίου αλλά με μεγαλύτερη επιμέλεια και σε ευρύτερη κλίμακα. Υπάρχουν διάφοροι νομικοί, δικηγόροι Φερρυπίν, που λένε ότι στο γαλλικό δίκαιο Φερρυπίν υπάρχουν όλα τα απαραίτητα μέτρα και δεν χρειάζεται ένα ειδικό νομοθετικό κόρπους για τα θύματα των επιθέσεων. Άλλοι όμως λένε ότι έστω και για όρους πολιτικής αναγνώρισης πρέπει να προβλεφθεί ειδική νομοθεσία και η ειδική μεταχείριση. Εμείς σε αυτή την επιλογή προέβημε, ότι χρειάζεται δηλαδή ένα ιδιαίτερο καθεστώ. Και έτσι με την ε, πρόταση της 30ης Ιουνίου προτείνουμε ένα ειδικό καθεστώς για τα θύματα, μπορείτε να την μελετήσετε. Ε, και αυτό ως τελευταία λόγια του ΣΥΠΗΝ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και το πιστεύω ότι πρέπει να δουλέψουμε όχι μόνο ε, με, ανα, σκημένη πάνω στο πρόβλημα, αλλά και με το κεφάλι ψηλά, το κεφάλι ψηλά στο όνομα της δημοκρατίας. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ Ζακτουμπό για την ώρα που μας χαρίσατε, για την έμφαση και την παρουσία με την οποία τοποθετηθήκατε μέσα από τις και την θέση που εκπροσωπείται και το θεσμό που εκπροσωπείται. Βέβαια ήξεραν οι συναδέλφοι ότι θα ερχόταν ε, ε, διαρκώ στο προσκήνιο το παράδειγμα της Γαλλίας, το περίμεναν άλλωστε και το θεωρούν ενδιαφέρον και για τις δικές μας τις εργασίες. Τίποτα πια δεν θα είναι όπως παλιά, ναι, αλλά ακριβώς αυτό εξετάζει η δική μας Επιτροπή το πώς θα μπορέσουμε να αναπηδήσουμε, να σταθούμε στα πόδια μας, όπως είπατε κι εσείς. Με σημαία ευρωπαϊκή, με τις δυσκολίες, τις νομικές, με τις δυσκολίες ως προς την εκτέλεση των κρατικών εξουσιών και των λοιπών αρμοδιοτήτων Και νομίζω ότι αυτό περιμένουν από εμά ε, του ευρωβουλευτέ ή πολίτε. Μια απάντηση ευρωπαϊκή, τουλάχιστον συντονισμένη σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και για τα θύματα. Επομένω και με τι βέλτιστε πρακτικέ ή τα βέλτιστα παραδείγματα ή τα υποδείγματα, αλλά και ως προς τη νομοθεσία που θα εισαχθεί. Και σε αυτό νομίζω δώσατε απαντήσεις ουσιαστικές και υλικό για μελέτη για την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και βεβαίως λέει ο κύριος Τουμπον, ε, είμαι εδώ παρόν με τους τρεις συνεργάτητες, τη Διευθυντρία καταρχάς, ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι με τις εργασίες του Κοινοβουλίου σας και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Εάν έχετε κάποια ερώτηση, κάποιο έγγραφο χρειάζεστε ή οτιδήποτε άλλο, είτε μέσω της Επιτροπής είτε απευθείας ε, ως μεμονωμένοι βουλευτές, ε, μην διστάσετε να μας ε, ζητήσετε πληροφορίες. Βεβαίως, λέει η Πρόεδρος, η Φχαυχώστε Σαμαρτά, η Μεριέλ Κουβέκ και η Κλοντίν Ζακόμπη, δική μας Κλοντίν, που έχει διευκολύνει τόσο πολύ την επικοινωνία με εσάς και έχει μακρά εμπειρία βέβαια από τα ευρωπαϊκά όργανα πριν έρθει στη δική σας υπηρεσία. Βεβαίως και περιμένουμε ότι θα υπάρχει συνέχεια στην συνεργασία μεταξύ των βουλευτών και της ομάδας σας. Σας εύχομαι καλή επάνωδο, πολύ καλές εργασίες. Ευχαριστούμε θερμά για την συνεργασία εδώ. Και υπενθύμιζω στους συναδέλφου ότι η προσεχή μα συνεδρίαση προβλέπεται για τις 22 Ιανουαρίου από τις 3 μέχρι τις 6.30 και την 3η 23 Ιανουαρίου από τις 9 έως τι 12.30 στι Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και καλή βραδιά σε όλου.